Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία ε, Ελίζα Φερέιρα, οριστήσα επίτροπο για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις. Καλωσορίζω επίσης ε, τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για συνδεδεμένες επιτροπές. Ενώ θέλω επίσης να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο που είναι παρόντες εδώ. Η ακρόαση αυτή αναμεταδίδεται και μάλιστα ζωντανά στο ιστότοπο του Κοινοβουλίου και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μάγνητο όπως προβλέπουν κατευθυντήριες γραμμές για την ε, έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράρτημα 7 του κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί τους οριστέντες επιτρόπους με βάση τις ε, γενικές ικανότητες, ε, την ευρωπαϊκή τους προσήλωση και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης αξιολογεί τη γνώση του μελλοντικού του χαρτοφυλακίου καθώς και τις ε, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν γύρε καμία ανιστάση ε, ως προς την διεξαγωγή της παρούσας ακρόασης. Ε, ήδη η οριστής Επιτρόπος έχει απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και οι γραπτές της απαντήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες στους βουλευτές της Επιτροπής μας. Καταρχάς τώρα να σας εξηγήσω πώς θα διαρθρωθεί αυτή η ακρόαση. Στην αρχή, στην αρχή συγγνώμη, καλείται η υποψήφια επίτροπος να προβεί σε μία εισαγωγική παρέμβαση, το πολύ 15 λεπτών. Εν συνεχεία, οι βουλευτές θα θέσουν 25 ερωτήσεις. Ο κάθε ένας θα έχει 5 λεπτά στη διάθεσή του. Ένα λεπτό για την ερώτηση. Δύο λεπτά η απάντηση της οριστίας σας επιτρόπου. Ένα λεπτό για επερώτηση στην οποία θα απαντήσει ξανά η Οριστής Επίτροπος μέσα σε ένα λεπτό το πολύ. Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα είναι από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και ο δεύτερος γύρος των 18 ερωτήσεων θα είναι σύμφωνα με την κατανομή των ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Θα υπάρχει και εκπρόσωπος από τους μη εργηγραμμένους συναδέλφους. Στο τέλος της συνεδρίασης θα δώσω το λόγο στην κυρία Φερέρα, οριστή σε επίτροπο για θέματα και μεταρρυθμίσεων και συνοχής για να προβεί σε μια καταληκτική δήλωση μέχρι στις διάρκειες 5 λεπτών και θα κλείσω εγώ για 3 λεπτά την συνεδρία. Είναι σημαντικό όλοι οι ομιλητές να σεβαστούν το χρόνο αγόρευσης για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεπεράσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και ορισμένοι βουλευτές δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Και όπως καταλαβαίνετε θα είναι πολύ ενοχλητικό κάτι τέτοιο. Όπως και στην Ολομέλεια λοιπόν θα υπάρχει χρονόμετρο που θα σας δείχνει το χρόνο και εφόσον τον ξεπεράσετε θα αναγκαστώ να κάνω χρήση του σφυρακίου που βλέπετε και να σας κόψω το μικρόφωνο. Κάτι το οποίο βέβαια ποτέ δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι και απαραίτητο δυστυχώς. Έχουμε στη διάθεσή μας διερμηνία σε 23 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μένους μπορούν να, να μιλήσουν στη μητρική τους γλώσσα. Όμως, ό,τι λέτε μεταφράζεται. Σας παρακαλώ λοιπόν να μιλάτε αργά για να διευκολύνετε το έργο των διερμηνέων. Κύριε Επίτροπε, κύριε υποψήφια Επίτροπε, πρωτού σας παραχωρήσω το λόγο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι προσεχής πέντε αιτία είναι πολύ κρίσιμη για το μέλλον της συνοχής. Διότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες, τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί με τις πολιτικές μας που κινητοποιούν πάνω από 350 δισεκατομμύρια στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού το 1 τρίτο δηλαδή του προϋπολογισμού της Ένωσης, παρόλα αυτά έχουμε κατακαιρματισμό και χάσμα μεταξύ των περιφερειών. Μέχρι τα τέλη του 2020 μας μένει Ενάμισης χρόνος για να αναδιαπραγματευτούμε τα πάντα και να καταλήξουμε σε συμφωνία πάνω ε, σε όλους τους κανονισμούς που αφορούν τη συνοχή. Μεταξύ αυτών έχουμε τον κοινό κανονισμό για όλα τα ταμεία, το ίντερεκ, το ΕΤΠΑ, το κοινωνικό ταμείο, ως παράδειγμα σας τα αναφέρω. Και πραγματικά ευελπιστώ να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο με τις διαπραγματεύσεις αυτές, να έχουμε λοιπόν ε, επικαιροποιημένους κανονισμούς, απλουστευμένους κανονισμούς, οι οποίοι όμως θα μπορέσουν να είναι πλήρως αποτελεσματικοί μόνο αν δεν μειωθεί ο προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και η Επιτροπή Προπολογισμών αγωνιζόμαστε για τον επαρκή προϋπολογισμό, για το προϋπολογισμό συνοχής στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το προσεχές πι. Υπάρχουν πολλές πιέσεις για μείωση του προϋπολογισμού της συνοχής, για την αντιμετώπιση νέων επιγουσών καταστάσεων. Πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία. Το χαρτοφυλάκιό σας περιλαμβάνει τη συνοχή και τις διδροτικές μεταρρυθμίσεις και αυτή η συσχέτιση είναι σημαντική και πρέπει να διασκεδαστούν οι ανησυχίες που μπορεί να προκύψουν. Κύριε Φερέιρα, χρειαζόμαστε στο πλευρό μας μία ισχυρή επίτροπο για τη συνοχή. Ισχυρή στο πλαίσιο του Σώματος των Ευρωπαϊκών Επιτρόπων για να μεταφέρει τις κοινέ μας φιλοδοξίες. να υπερασπιστεί τα άρθρα 174 και 175 σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω θα χρειαστούμε ε, μια επίτροπο η οποία θα ακούει την Επιτροπή Ρέγγι και σημειώνουμε την πρόταση της Πρόεδρου Φοντερ για την καθιέρωση ενός δικαιώματος πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν υπάρχει ένα κοινό όραμα, ένα κοινό σχέδιο, αν δεν ε, φιλοδοξούμε να υπάρχει μια ανάπτυξη ισορροπημένη και συνοχή σε όλες τις περιφέρειες, δεν πρόκειται να υπάρξει ένα κοινό μέλλον, ένα κοινό πεπρωμένο για όλη την Ευρώπη, διότι η συνοχή ε, σημαίνει ε, μια στροφή πολύ σημαντική και είναι το αντίδοτο σε οποιαδήποτε κρίση. Η ιδέα αλληλεγγύη είναι στον πυρήνα βέβαια. Η ακρόαση αυτή είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ επικοδομητική. Με τα χαράς λοιπόν κυρία Ελίζα Φερέρα σας δίνω τώρα το λόγο για 15 λεπτά. Πρωτού προχωρήσουμε στη συζήτηση με τα μέλη των επιτροπών μας. Merci, Monsieur le κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πρόκειται για μια φορτισμένη συναισθηματικά το να είμαι στην συνάντησή και πρόκειται για ε, τα αγγλικά τα οποία χρησιμοποιώ τώρα είναι γλώσσα εργασίας αλλά επίσης ε, ε, στα αγγλικά αν σας τα πω θα είναι απευθεία επικοινωνία. Θέλω να σας πω επομένω ότι εδώ πέρασα ένα σωρό χρόνια, 12 χρόνια εδώ στην καρδιά της Ευρώπης, πολύ καλή ανάμνηση και με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ε, εδώ ότι βρίσκονται από την Ρέτζη, από την ΕΚΟΝ, από την Επιτροπή των Προπολογισμών οι παλαιοί συνάδελφοι. Και σήμερα είναι τιμή μου να παρουσιάσω αυτή την πρόταση για την επόμενη πενταετία. Και ε, ως ε, παλαιά ευρωβουλευτής κατανοώ το πόσο σημαντικό είναι το έργο το οποίο επιτελείται και πραγματικά πιστεύω ότι μόνο ε, αν προχωρήσουμε χέρι-χέρι μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη, να υπάρξει ελπίδα για το ευρωπαϊκό όραμα από όλους τους Ευρωπαίους όπου και να βρίσκονται εκείνοι. Η κυρία Κρέτσου, η προκατοχός μου, αξίζει συγχαρητηρίων, δεν άφησε καμία περιφέρεια στο περιθώριο και εγώ θα προσθέσω να κάνω το ίδιο και να προσθέσω και την προσωπική μου εμπειρία. Ε, καμία περιφέρεια στο περιθώριο. Να, τι θέλουμε. Για την ψηφιοποίηση, για την αλλαγή του κλίματος, για, για τα πάντα. Θα πρέπει κανείς να μην χάσει το τρένο και θα πρέπει να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν για το μέλλον. Θα βεβαίω η αλλαγή δεν και το έχω διαπιστώσει και προσωπικά Είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα πλαίσιο, ήταν ε, δύσκολα για την κλωστοφαντουργία ε, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τις ε, κοινότητες και τους δήμους που εξαρτιόντουσαν οικονομικά και πάρα πολύ πρόσφατα διπιστώσαμε τι έγινε στο, στην, με το στον απόϊχο της κρίσης του 8 διάφορες βιομηχανίες, διάφορες μέρη αλλά με το ίδιο σενάριο και δε ποτέ δεν ξεχνούμε τα κλειστά εργοστάσια, τους ε, εργαζόμενους στον δρόμο, ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ε, μείωση των ε, μισθών και κυρίως τους νέους, τους ευφυείς νέους, τους ικανούς που φεύγουν για το εξωτερικό, αλλά χρειάζεται μια μεταρρύθμιση, χρειάζεται να υπάρχει και συνοχή. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας οι κορυφαίες και έχουμε παγκοσμιοποίηση, έχουμε τεχνολογική επανάσταση, όλα αυτά πιέζουν πάρα πολύ τις οικονομίες κάθε τόπου. Και πιστεύω στην περιφερειακή πολιτική γιατί έχω δει τις επιπτώσεις της επιτόπου και από τότε που ήμουν νέο οικονομολόγος σε θέματα ανάπτυξης ή υπουργό ε, προγραμματισμού και χρωταξίας είδα ότι είναι μοχλός αλλαγή στην Ευρώπη αυτή η υπόθεση και χρωταξιας ειδα οτι ειναι μοχλος αλλαγη στην ευρωπη αυτη η υποθεση για κάποιες περιφέρειες είναι το μόνο μέσο που υπάρχει από την Αρκτική στην Μεσόγειο, από τις ε, πόλεις σε αποβημενισμένες περιοχές μέχρι δηλαδή ε, την απότερη περιφέρεια της Ένωσης από τα βουνά μέχρι την ε, Ήπεθρο από τις περιφερειακές ε, παράλληλες περιοχές μέχρι τα σύνορα θα πρέπει όλα αυτά να απασχολούν την Ευρώπη θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και οι Ευρωπαίοι μια οικονομία για τον άνθρωπο με κάποια ε, μέσα οικονομικής πολιτικής στα μέτρα του κάθε τόπου να βάλουμε υπόψη την ισότητα των φύλων, την την τεχνολογία, την, την διάσταση περιβάλλον. Οπότε, αγαπητοί βουλευτέ, είναι τιμή μου που αναβάνω αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και η κυρία Φόντερ Λάιεν, η νεοκλέξα πρόεδρος, ε, μα είπε ότι μας έδωσε ε, ε, κάποια καθήκοντα πολύ σημαντικά. Πρώτα-πρώτα το νομοθετικό πλαίσιο και μας τόνιζε και συμφωνώ μαζί της ότι χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία ταχείας και έτσι να αρχίζουν να τρέχουν ε, προγράμματα από την πρώτη μέρα καθήκοντων μας. Και εγώ ποντάρω σε εσά, στη συνεργασία μαζί σας. Να υπήρχε επίσης το Ταμείο για την Μετάβαση μεταβατική περίοδο και έχω ήδη προτείνει να στριχτούν οι περιοχές εκεί που υπάρχουν οι μεγάλες προκλήσεις κυρίως ε, από πλευράς βιομηχανίας, από πλευράς ε, έντασης εργασίας, ε, όπου χρησιμοποιείται άνθρακας και όλα αυτά θα αποτελούν την Επιτροπή της πρώτης 100 μέρες των καθηγόντων επίσης να γίνει ομαλή εφαρμογή επομένως το, στην επιστολή μου τα λέω ξεκάθαρα θα πρέπει η πολιτική να είναι σύγχρονη, απλή για να πάει σε ποιοτικέ επενδύσεις να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη στενά, απλούστευση ε, τέρμα στη γραφειοκρατία να υπάρχουν όμως ποιοτικοί έλεγχοι και προγράμματα με διαχείριση υγεία και αυτά να έχουν το ρόλο τους με επιπτώσεις θετικές και όσο γίνεται να υπάρχουν συνέργειες με την πολιτική συνοχή. Οι προτάσεις μας είναι φιλόδοξες. Για παράδειγμα θέλουμε η cost το κόστος να πλουστεύεται στις επιλογές μας και επίσης να έχουμε 25% μείωση ε, του κόστους γραφειοκρατίας και θα πρέπει να ελέγχετε κατά πόσον οι εξαγγελίες μας υλοποιούνται. Θεωρούμε ότι εσείς είσαστε σύμμαχοι σε όλα αυτά, στην προσπάθεια δηλαδή της απλούστευσης ε, τρίτο θέμα χαρτοφυλακείο, οι μεταρρυθμίσεις, η νομισματική ένωση είναι μια πρόκληση, αλλά ε, η αντιγωνιστικότητα έχει κάθε χώρα. Ιδίω δε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετική συγκυρία ε, και κοινωνικές συνθήκες που να είναι βιώσιμη η αλλαγή, ανταγωνιστικότητα να είναι το θεμέλιο σε αυτή την προσπάθεια επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικά και για αυτό ήρθε η ώρα να ξαναρχίσει η συζήτηση για νέα υποστήριξη των επενδύσεων. Να υπάρχει αντιστοιχό πρόγραμμα και να βοηθήσει και ο προπολογισμό για σύγκληση και αγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη. Το ευρώ είναι το νόμισμά μας και θα πρέπει επομένως έγκυρα να υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές που ήδη έχουν μπει στην Ευρωζώνη. Επίσης και εκείνους που κάνουν σοβαρές προσπάθειες προς τούτο η μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αυθυγραμμίζονται και με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Επίσης θα πρέπει όλα να περνάνε από την έγκριση της χώρας που εμπλέκεται να μην μπλοκάρεται πουθενά η βιώσιμη ανάπτυξη, σύγκληση, ανταγωνιστικότητα σημαντική, βοήθεια στα εθνικά προγράμματα και να εξυγχρονίζεται η δημόσια διοίκηση και ε, να βελτιώνονται και η διαχείριση των δασών, ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε το ένα όργανο τον άλλο. Οι δε φορολογούμενοι να μην ε, χρηματολογούν, μην χρηματοδοτούν κάποιες ε, πολιτικές που δεν όφελουν. Ε, Στενή σχέση με το Κοινοβούλιο, γιατί με τέτοια μέσα πολιτική θα προχωρήσουμε με την κοινοτική μέθοδο. Είναι σημαντική η δική σας βοήθεια και έτσι θα έχουμε πρόοδο. Έτσι θα μπορέσουμε να κινηθούμε στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται. Βιώσιμη ανάπτυξη υπαίθρου και πόλεων. Πρόκειται να γίνει αναθεώρηση του θεματολογίου και η πόλη σήμερα είναι αιστεία κακής στέγασης, φτώχειας, ανεπαρκών μεταφορών, βλάβης του περιβάλλοντος και όμως έχουμε και ευκαιρία μέσω των πόλεων. Οι πόλει μπορεί να είναι πρωτοπόρε για την πράσινη οικονομία, την ψηφιακή οικονομία. Υπάρχουν ευκαιρίες, α εκμεταλλευτούμε στενή συνεργασία με τις τοπικές ε, αρχές. Στο Πόρτο, τον Ιανουάριο του 20 θα κάνουμε ένα φόρουμ για τις πόλεις. Θα είναι ευτύχημα αν έρθετε. Επίσης, την απότερη περιφέρεια να φροντίσουμε. Το λέει και η συνθήκη και έχω αναγνωρίσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένε ε, ανάγκε. Χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Επίση, ε, οι περιοχέ που είναι κοντά στα σύνορα και οι ορεινέ. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό ότι η διάσταση αυτή έχει καλυφθεί από 21 διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις από αελεία μέχρι έρευνα, μέχρι αλλαγή του κλίματος και μεταφορές και ήδη αυτά έχουν περάσει από ένα τεμερή διάλογο, άλλες προτάσεις θα πρέπει να τις προωθήσουμε, όλα αυτά μαζί σας. Επίσης, έκτο και τελευταίο τμήμα είναι η επικοινωνία, πρόκειται για κάτι που έχει σημασία για πάρα πολύ κόσμο, ακόμα δεν κάνουμε αρκετά και αυτό που θέλω είναι να πάω παντού, να καταλάβω τον προβληματισμό, να δω τι εμπνέει τον κόσμο και έτσι να υπάρχει καλύτερη υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων και κανείς να μην φοβάται ότι έχασε το τρένο, τον αφήσαμε πίσω και γι' αυτό και πάντοτε θα σας ενημερώνω όποτε πάω στο δικό σας τόπο και θα σας λέω τις πρωτοβουλίες μου και θέλω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω με τις επιτροπές που σήμερα εκπροσωπούνται εδώ προτεραιότητα για την πρόεδρό μας αλλά και για μένα την ίδια. Σας είπα ποια είναι η αποστολή μου και κλείδι να σας πω δύο λόγια για τον εαυτό μου, να σας πω εγώ πώς θα συμβάλλω σε όλα αυτά πρώτα-πρώτα. Πραγματικά πιστεύω σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και υπόσχομαι ότι θα ε, αποδώσει και έχω προσωπική εμπλοκή και ενδιαφέρον γιατί κάθε μέρα της ζωής μου ξέρω τι γίνεται με αυτή την πολιτική. Έχω ακούσει πάρα πολλά για το τι σημαίνει μεταρρύθμιση, τι σημαίνει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και είχα εργαστεί ως οικονομολόγος επί τόπου. Είδα το πόσο πιάνει τόπο αυτή η πολιτική στην καθημερινή ζωή. Ήμουνα υπουργό πρόσφατα για την πολεοδομία, τη χωροταξία ε, και είχα συμβάλει στην ε, επιτυχία του προγράμματος πλαισίου 2000 μέχρι το 2006 και ε, που λαμβάνω απόψη και το έργο του κυρίου Μπαρνιέ και επίσης είχα εργαστεί στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Κεντρική Τράπεζα ως ε, ε, διοικητής στη χώρα μου και έμαθα τα οικονομικά κατάλαβα γιατί λέγανε ανέκαθεν ότι η συνοχή και η ανταγωνιστικότητα είναι κλειδιά της αποτυχίας οπότε από τα πανεπιστήμια μέχρι τη δουλειά μου, μέχρι την τράπεζα, στο κοινοβούλιο, όλα αυτά τα επιστράτευσα και οπότε θα πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο. Ότι εγώ είμαι ο παδός της ομαδικής προσπάθειας, θα συνεργαστώ και στην Κομισιόν και με εσά και με τον ντόπιο κόσμο και με τις, και με τις κοινότητες και τους δήμους και επίσης νομίζω ότι για πρώτη φορά υπάρχει ισορροπία των δύο φίλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ επίσης είμαι η πρώτη από πλευράς Πορτογαλίας που συμμετέχει άρα θα πρέπει να σπάσουμε τα στεγανά να έχουν οι γυναίκες ε, ε, το, το πιδάλιο στα χέρια τους και θα γράψουμε πάνω στην ιστορία όντας περήφανοι γι' αυτό και εν κατακλείδη πιστεύω στην Ευρώπη μας. Αυτά ε, πολύ πριν αρχίσω να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο την ε, ολοκλήρωση. Ο Βίλ Μπραντ, ο παλιός καγκελάριος, ήταν πολύ σπουδαίος ε, και ε, θυμάμαι ότι μεγάλωσα σε μια δημοκρατία, αλλά η Ευρώπη έφερε την δημοκρατία. Όπως και ο Μάριο Σουάρες, θέλω μια ελεύθερη Πορτογαλία στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Να, τι σημαίνει για μένα Ευρώπη ίσον δημοκρατία και βλέποντας επί τόπου κατάλαβα τι σημαίνει αλληλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία όταν κανείς δεν έχει υγεία, παιδεία, κοινωνική πολιτική άρα Ευρώπη ίσον αλληλεγγύη για μένα και όταν έγινε να κατάλαβα ότι σημαίνει και φιλία, αλληλοσεβασμό, κοινέ αξίες και αυτό το ενωμένη στην πολυμορφία. Άρα όλα αυτά και ακόμα περισσότερα πάει να πει η Ευρώπη για μένα σήμερα, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Ευρώπη Δημοκρατία, αλληλεγγύη, φιλία, κοινών αξιών μέσα στην πολυμορφία. αυτή η Ευρώπη μα στέλνει μήνυμα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τα ψηφιακά, την ψηφιακή εποχή, την ψηφιακή οικονομία, η Ευρώπη απαιτεί να δείξουμε τόλμη, τόλμη να προωθήσουμε την συνοχή και την μεταρρύθμιση. Και έτσι κανένα, καμιά περιφέρεια να μην μείνει πίσω. Άρα, σε αυτό το κάλεσμα τη Ευρώπη, θα σας απαντήσουμε όλοι μαζί, κύριε Πρόεδρε, στα γαλλικά. Αυτό θα κάνω εγώ. Θα απαντήσω αυτό το κάλεσμα γιατί έχω το, την, την, την τιμή να υποβάλω την υποψηφιότητά μου ω επίτροπο για μεταρρυθμίσεις και συνοχή. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσει σας και σα ευχαριστώ και στα πορτογαλικά. Madame Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φερέρια διότι ήσασταν άψογοι με το χρόνο Τον τηρήσατε απόλυτα, οπότε μπορεί τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε καταρχά τον πρώτο γύρο με του συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι έχουμε τα πεντάλεπτα όπως σας είπα, δηλαδή ερώτηση ένα λεπτό, απάντηση δύο λεπτά, επερώτηση δεύτερη ένα λεπτό και απάντηση δεύτερη άλλο ένα λεπτό. Πρώτος το λόγο έχει ο συνάδελφός μας από το ΕΛΚ, Αντρέι Νοβάκοφ. Dear Commissioner Designate, I feel proud today υποψήφια επιτροπέ. Είμαι περήφανο σήμερα γιατί αντιμετωπίζετε την ομάδα του ΕΛΚ η οποία αντιστάθηκε όταν όλοι οι άλλοι ήθελαν περικοπές στην πολιτική συνοχή. Η ομάδα αυτή μαζί με τις άλλες πολιτικές ομάδες είναι ακριβώς αυτή η οποία υποστήριξε την στεναρή θέση του Κοινοβουλίου για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η ίδια αυτή ομάδα μας έδωσε μία εντολή πριν από λίγες ώρες να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει για το μέλλον αυτή τη πολιτική. Γι' αυτό σα ερωτώ, θα στηρίξετε αυτή την ομάδα και την θέση του Κοινοβουλίου για να στηρίξουμε τον προπολογισμό τη συνοχή ή θεωρείτε ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τη συνοχή και θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές. Θα συμφωνήσετε στην ανάκτηση του ποσοστού συγχρηματοδότηση για τι φτωχότερε περιοχέ ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Νοβακόφ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί θα με βοηθήσει να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι η πρόταση που παρουσίασε η Κομισιόν είναι απλά μια βάση, μια αφετηρία. Μια αφετηρία η οποία περιλαμβάνει διάφορα ζητήματα, τα οποία είναι θετικά και επαρκή. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ένας περιορισμός. Όταν ε, συζητάμε εμείς τον προπολογισμό αποφασίζουμε μόνο τις δαπάνες ε, και όχι τα εισοδήματα. Αυτά τα αποφασίζετε εσείς και τα κράτη-μέλη. Οπότε, οι δύο συνομοθέτες μεταξύ σας θα αποφασίσετε ποιο θα είναι το ύψος του προϋπολογισμού. Οπότε, εγώ, στην Κομισιόν και οπουδήποτε αλλού, θα στηρίξω οπωσδήποτε το θέμα αυτό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Όχι απλά επειδή είμαι υποψήφια για αυτή τη θέση, αλλά επειδή πραγματικά πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εμβαθυνθεί, να διευρυνθεί και να συνεχίσει να έχει περιορισμένα κονδύλια. Βεβαίω το τελικό αποτέλεσμα θα είναι περιορισμένο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση αυτής της ε, πολιτικής και στο πώς ε, αναλύουμε τον χωρικό αντίκτυπο των ε, τομεακών πολιτικών. Αλλά οπωσδήποτε εντό του πλαισίου ελιγμών που έχουμε θα κάνω ό,τι μπορώ απέναντι στους άλλους συναδέλφους μου για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο χρηματοδότησης για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, συμφωνώ ότι Ακριβώς η πολιτική συνοχής είναι η συγκολητική ουσία της Ένωση, αλλά είμαι σίγουρο ότι κανείς έξω από αυτήν την αίθουσα δεν αντιλαμβάνεται γιατί εφαρμόζεται τόσο αργά. Οπότε, πώς σκοπεύετε να αποφύγετε την καθυστερημένη εφαρμογή αυτή τη πολιτική έχοντας κατά νου ότι ένα έτος πριν από το τέλος της προγραμματικής περίοδου η εφαρμογή είναι μόλις στο 30%. Νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε το ποια είναι τα μυστικά ε, των ε, δικαιούχων, με τι πρέπει να συμμορφωθούν για να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια. Με βάση αυτό η τωρινή πρόταση της Κομισιόν είναι πολύ σαφής. Ε, η απλοποίηση είναι στο επίκεντρο της ατζέντα μας. Υπάρχουν πάνω από 80 προτάσεις που βρίσκουν και το Κοινοβούλιο σύμφωνο. Ελπίζω λοιπόν στο Συμβούλιο να έχουμε αυτήν την ε, συναντήληψη. Ο στόχος πολιτικής είναι να έχει αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ξεκάθαρα το αν υπάρχουν κάποια εμπόδια στην αποτελεσματικότητα οπωσδήποτε πρέπει να επιταχύνουμε έτσι ώστε ο κόσμος να νιώσει επιτόπου τον αντίκτυπο αυτής της προσπάθειας που κάνουμε έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να εργαστεί όχι κατακαιρματισμένη αλλά πιο ενωμένοι έτσι ώστε όλοι οι πολίτες όπου και αν βρίσκονται να νιώθουν μέρος αυτού του εγχειρήματος. Αυτός είναι ο στόχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές τον λόγο έχει η συνάδελφός μας κυρία Κωνσταντς Κρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Φερέρα, αγαπητή Ελίζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ε, προκλήσεις. Παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, κλιματική αλλαγή, δημιουργία καλών θέσεων εργασίας και τα λοιπά. Πώς μπορεί να συνεισφέρει λοιπόν η πολιτική συνοχής για να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των περιοχών και να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Αγαπητή κυρία ε, βουλευτή, τι, κυρία Κωνσταντίνος. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η πολιτική θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Θα επιταχύνουμε την σύγκληση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα κονδύλια που έχουμε. Τα κονδύλια αυτά βεβαίως ε, ελπίζω να αυξηθούν, αλλά είναι περιορισμένα. Πάντα έχουμε καινούργια θέματα ε, και ο γενικός φάκελος σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε το τι θα κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Πράσινη μετάβαση, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, νέα κοινωνία Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στις περιοχές που χρειάζονται τα κονδύλια περισσότερο, να δούμε τις φτωχότερες περιφέρειες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες και στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ε, ξόχως ε, απομακρυσμένες και πρέπει να δούμε τις περιφέρειες εκείνες που είναι σε μετάβαση ίσως να ήταν πολύ βιομηχανοποιημένες ε, και τώρα να αντιμετωπίζουν μια κρίση. Πρέπει να μετασχηματίσουν το μοντέλο τους και πρέπει να σχηματίσουμε ένα πακέτο για αυτές τις ε, περιοχές, ε, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώνται από την βαριά βιομηχανία ή το λιγνίτη ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που ακριβώς αυτό το ζήτημα θα αντιμετωπίσει. Πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα μέσα μας στα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας. Να υπάρχει μια ευελιξία που θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την διαδικασία σύγκλησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να συνεισφέρει η πολιτική συνοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα μέλλον ουδέτερο ως προς τις εκπομπές. Και πώς βλέπετε την πολιτική αυτή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Green New Deal. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν συμβιβασμό σε σχέση με το Περιφερειακό Ταμείο ότι 30% των πληρωμών στην επόμενη περίοδο 2021-2027 θα πάει προς ε, έργα κλιματικά ανταγωνιστικά και το κατόφλι είναι υψηλότερο, είναι 37% για το Ταμείο Συνοχής, δεδομένου του ότι αυτά τα δύο ταμεία προσωπεύουν το 35% του κοινοτικού προπολογισμού και 25% και μαζί με το άλλο ταμείο είναι ένα τρίτο του προπολογισμού. Ε, θα δώσουν νομίζω μια νέα όθηση προς ε, μια πιο γρήγορη συμμόρφωση της ε, Ευρώπης με τους κλιματικούς στόχους. Στο παρελθόν είχαμε κάποιες προσπάθειες, 25% του προηγούμενου πακέτου είχε αφιερωθεί σε έργα που αφορούν το κλίμα. Τώρα έχει αυξηθεί και επιπλέον έχουμε διάφορες γραμμές ε, του προϋπολογισμού που μπορούν να συνδυαστούν για να εκμεταλλευτούμε πλήρως το κλιματικό πακέτο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ομάδα Renew. Το λόγο έχει στον Άφης Αντρέη Κνότεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρία Φερέρα. Έχω μια ερώτηση για το Ταμείο Δικές Μετάβασης, που είναι ένα βασικό εργαλείο για την μετάβαση μια χαμηλών εκπομπών ε, οικονομία. Αυτό το ταμείο πώς ε, θα το σχεδιάσετε, τι χρηματοδότηση θα έχει και ποια θα είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, για τα έργα και τις περιφέρειες που θα υποστηρίζει και όπως και με την πρόταση για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, υπάρχουν και εδώ προτάσεις για Μάλλον υπάρχουν προτάσεις για περικοπές, αλλά δεν περιλαμβάνεται το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Θα προσπαθήσετε να υπάρξει εγγύηση ή κάποια άλλη δέσμευση ότι δεν θα περικοπούν ε, τα κονδύλια ε, για αυτό το Ταμείο βάζοντας μεγαλύτερη πίεση ε, σε αυτή την πολιτική απάντηση. Αγαπητέ είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σα, διότι αυτό το Ταμείο Δίκαιες Μετάβασης η κυρία Φοντρελάιν το έχει ε, θεωρήσει ένα σύμβολο για την Επιτροπή της. Ε, ήταν ε, κάτι που ξεκίνησε από το Κοινοβούλιο το 2018. Ήταν δικό σας αίτημα, να μην το ξεχνάμε, και με ψήφισμά σας και ένας από τους συνεισηγητές είναι εδώ, η συγκεκριμένα η κυρία Καρδιά Θάμπαλα που ζητούσε και επικοδότησε ακόμα Το κοινοβούλιο βέβαια ζητούσε τότε 1,3% του καθάριστου εθνικού σοδήματος. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να υποσχεθώ είναι πως το ταμείο αυτό θα λειτουργήσει, θα συνεχίσουμε το προπαρασκευαστικό έργο ε, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί προς το παρόν είμαστε όλοι υποψήφοι. Θέλουμε να δοθεί όμως μια ε, τοπική προσαρμοσμένη στις ανάγκες υποστήριξη. Θέλουμε να προωθήσουμε επενδύσεις με στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης για να έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, ένα νέο παράδειγμα σε σχέση και με την κλιματική αλλαγή το περιβάλλον. Θέλουμε να είναι πιο βιώσιμο για το μέλλον. Ταυτόχρονα Μελετούμε όλες τις λεπτομέρειες για να δούμε πού θα προέλθει η χρηματοδότηση του Ταμείου. Θα συνεργαστώ στενά με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο για την πράσινη με τον Επιτρόπο για την Ενέργεια, για τη διαχείριση του προπολογισμού. Βέβαια, ειλικρινά σας το λέω, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξέρουμε από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Εγώ θα προτιμούσα να συμπληρωθεί αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με νοπό χρήμα. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω υποσχέσεις αυτή τη στιγμή. Ξακολουθούμε αυτή τη στιγμή να εργαζόμαστε πάνω στο συνολικό πλαίσιο και έπειτα θα δούμε πώς θα οργανώσουμε τη χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού που σίγουρα θα συσταθεί και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιφέρειες που εξαρτώνται από τη βιομηχανία, από την ενεργική κατανάλωση, τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο συγκεκριμένα για τις ε, περιοχές ε, με πολλά ανθακοριχεία, Ιδίω αυτέ θα επηρεαστούν από τη μετάβαση με οικονομία χαμηλών πομπών άνθρακα και χρήση άνθρακα. Πώ βλέπετε αυτέ τι περιφέρειε, ε, τι ρόλο έχουν ω δικαιούχοι του Ταμείου Δική Μετάβαση, θα είναι πράγματι οι βασικοί δικαιούχοι. Απάντηση. Ο λόγο ύπαρξη του Ταμείου δικαιοσύνη μετάβαση είναι ακριβώ να ανταποκριθεί στις πολύπλοκε αυτέ καταστάσει πώ θα οργανώσουμε τη μετάβαση που είπατε. Σε συνδυασμό με τα Ταμεία συνοχή και τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν, θέλουμε επιτόπου σε τοπικό επίπεδο να προσπαθήσουμε οι περιφέρειε αυτέ να ε, αλλάξουν εντελώ να διαρθρωθούν. Θέλουμε ένα νέο παράδειγμα που σα είπα. Δεν μπορώ να σα πω αν θα είναι οι μόνε δικαιούχοι. Θα αναλύσουμε με μεγάλη προσοχή και όλες τις άλλες ε, περιφέρειες που ενδεχομένω χρειαστούν υποστήριξη. Ο στόχο είναι όμως ε, να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές να ανακτήσουν το χαμένο έδαφο ε, και να ξεφορτωθούν αυτό το βάρος, αν θέλετε, που είναι ένα βάρος για όλη την Ευρώπη και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τώρα τον αγαπητό συνάδελφο Νίκλα Νίνας να κάνει τι ερωτήσει του εκ μέρου της ομάδας των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Κύριε Φεραίρα, χαίρομαι ιδιαίτερα που η κλιματική αλλαγή είναι μείζον ζήτημα για την Επιτροπευτή και θέλω να κάνω μια ερώτηση για την κλιματική αλλαγή, διότι αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο ω Ευρωπαίοι, αλλά ω ανθρωπότητα εν γέννη. Χρειάζεται λοιπόν άμεση δράση. Είδαμε λοιπόν οι νέοι Ευρωπαίοι να κατεβαίνουν στους δρόμους και να διαδηλώνουν. Είδαμε και στην προεκλογική εκστρατεία ε, να είναι ένα από τα θέματα κλιματικά που μονοπολούσε. Ε, μόνος χρειάζεται ε, δράση, είπε η κυρία Φοντρελάιν, ακολουθώντα το το κλίμα αυτό, ότι θέλει να μειωθούν μέχρι το 2030 κατά 55% οι εκπομπέ των κυπριακών αερίων η συνοχή θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Το 50% νομίζω των ε, δαπανών του θα πρέπει να αφαιρωθεί ακριβώ σε αυτό το στόχο, το μετρησμό τη κλιματική αλλαγή. Θα φροντίσετε να επιτευχθεί ο στόχο αυτό, αυξάνοντα τουλάχιστον το 5% τη δαπάνη για το κλίμα. Θα αγωνιστείτε για την ε, καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών για κλιματικέ ενέργειε ε, σε επίπεδο τμήματων και διευθύνσεων και τη Γενική Διευθυνσή σα. Πώ θα επιτύχουμε πρόοδο για την <clears throat> μείωση ε, της χρήσης άνθρακα. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ σοβαρό το ερώτημα, διότι η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγή ε, δεν μπορεί να είναι κατακαιρματισμένη, πρέπει να είναι οριζόντια και πρέπει να ενσωματωθεί σε όλε τι πολιτικέ. Νομίζω ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως ο συμβιβασμό ε, της Προέδρου Φοντρι ε, και η δέσμευσή της μάλλον είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια θα πρέπει να πολύ συγκεκριμένοι για να οργανώσουμε με πολύ προσεκτικό τρόπο τα διάφορα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε δει το στόχο για το 2030 και έχουμε και το στόχο για το 2050. Αυτό ζητά, απαιτεί τεράστιες μαζικές επενδύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο την πολιτική συνοχή που είναι και το βέβαιο και έχουμε και τα κατόφλια αναπεριφέρεια 30-60% ανάλογα με το επίπεδο των περιφερειών και χωρών, μιλάω για το επίπεδο ανάπτυξης. Και έπειτα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Τάμιο Καινοτομία, ε, το ETS, ε, με το Horizon Ευρώπη, την ε, ανακατανομή κονδυλίων των υφιστάμενων εργαλείων, το InvestEU, το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή συνδυασμένα. Έχουμε πολλά, το IP και όλα αυτά τα εργαλεία, για να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα με στόχο να πετύχουμε όλα αυτά που ξέρουμε ότι θα είναι δαπανηρά και τεχνικώς πώς δύσκολα να επιτευχθούν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το σωστό ε, δρόμο, ε, να επιταχύνουμε, να βρούμε τη σωστή ταχύτητα, σωστό ρυθμό. Αλλά σίγουρα αυτό είναι ο στόχος αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριος ε, Νίνας. Σας ευχαριστώ. Οι περιφέρειες οι οποίες τώρα βασίζονται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες ε, μετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για να διατηρήσουν αποδεκτά ε, συνθήκες διαβίωσης. στις περιοχές ε, με ανθακοριχεία, στις περιοχές ε, της ενεργοβόρης βιομηχανίας ε, θα εστιάσουμε. Θέλουμε όμως να προετοιμάσουμε για το μέλλον της περιφέρειας, αν δεν θέλουμε άνθρακα. Θέλουμε 100% απαλλαγή από άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις περιφέρειες για να μετασχηματιστούν. Εδώ περιλαμβάνεται οικονομική και κοινωνική διάσταση. Πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό είναι μείζονο σημασία. Στηρίζεται την απόσυρση μέχρι το 2030 από, την, ε, από τον άνθρακα, όπως απαιτεί η Συμφωνία των Παρισίων και πώς θα περιλαμβάνεται στο JTF η καταπολέμηση της φτώχειας και επειδή μίλησαν για τη χρηματοδότηση συνάδελφοι, θα πρέπει να γίνει εσωτερήκευση ε, του εξωτερικού κόστους ε, για το JTF, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. In a, very short, ε, Να σας τα πω τηλεγραφικά. Σίγουρα πρέπει να το ψάξουμε, να δούμε πώς το ETS θα χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό και επίσης να δούμε και τα προγράμματα αυτών των προγραμμάτων τα οποία δεν μπορεί να αποδώσουν ή αν δεν συνδυάζουν τον κοινωνικό παράγοντα, τον επενδυτικό, αλλά και την οικονομική πτυχή. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να συγκεραστούν για να αποδώσει το πρόγραμμα. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να συνεργαστούν σε τοπική κλίμακα και να μην ξεχάσουμε να συνδυάσουμε και το Ταμείο της Μετάβασης. Με τον πέμπτο στόχο δηλαδή. Το πώς ολοκληρωμένα όλα αυτά θα συνδυαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια βάση της πολιτικής και των κατευθυντηρίων. Άρα συνέργεια και προσπάθεια για βιωσιμότητα. Ε, συμφωνούμε 1000%. Je cède la parole à Francesca Donato. Francesca Donato, Να σας τα πω στα Ιταλικά, Πρόεδρε, λέει η κυρία Ντονάτ. Ευχαριστώ, κύριε υποψηφία Επιτροπέ. Μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχετε ανοιχτό πνεύμα και πρόθεση συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και σας ερωτώ, η Επιτροπή προβλέπει μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η κρίση δικαιολογούσε τα υψηλά ποσοστά και θεωρείται ότι τέλειωσε η κρίση. Αλλά έχουμε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές όπω στο νότιο τη Ιταλία, κάποια νησιά και εκεί επιβάλλεται στήριξη. Χρειάζονται αυτά τα ταμεία και τα κονδύλια. Οπότε λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα, ευελιξία του ποσοστού. Να ληφθεί υπόψη η κοινωνική συγκυρία, η οικονομική συγκυρία του κάθε μέρους. Σας ευχαριστώ και θεωρώ ότι, λέει η κυρία Επίτροπος, το θέμα της ανάπτυξης της Νοτιού Ιταλίας θα πρέπει να εξεταστεί. Αποτελεί ένα μάθημα το πώς μπορούμε να δώσουμε δυναμισμό σε μια περιοχή γεμάτη προβλήματα. Μας δώσετε ένα παράδειγμα. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε το πόσο χρειάζεται να έχουμε θεσμούς ισχυρούς κατάλληλη διαχείριση των αντιορθωτικών ταμείων, ανάλυση των δεδομένων και λήψη αποφασιών. Επίσης, να μην ξεχνούμε τις ιδιορυθμίες και ιδιοτυπίες κάθε μέρους και των λοιπόν εμπλεκομένων. Και φυσικά για το ποσοστό τη χρηματοδότηση θα ξέρετε το 2009 οι ποσοστώσεις, τα ποσοστά τέλο πάντων, ευξήθησαν. Δηλαδή βοηθάγε περισσότερο η Ένωση τα εθνικά προγράμματα. Είχαμε τα προβλήματα βέβαια της κρίσης από το 8 και αυτό ήταν το θέμα. Οπότε θα πρέπει να γίνει κάποια παρέμβαση αντικυκλική. Και έτσι να αντισταθμίσουν τα προβλήματα σε επενδύσεις και θα πρέπει να γυρίσουμε στην ε, κανονικότητα. Και αυτό όμως με προσοχή. Δεν θα πρέπει να βιαστούμε. Να μην αλλάξουμε το ποσοστό τη συγχρηματοδότηση χωρί να ξέρουμε τι επιπτώσει θα υπάρχουν. Πάντω, ε, αυτή είναι η ρότα που θα πάρουμε. Επιρώτηση κυρία Ντονάτο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ρωτώ, όσον αφορά αυτό του είδους ε, τις περικοπές στο πρόγραμμα πλαίσιο για συνοχή και για ΚΑΠ, εσείς υπόσχεστε να φρενάρετε κάποιο είδους μετακίνηση ή περικοπής αυτών των ε, κονδυλίων. Για να μην γίνει η σχετική πολιτική σε σχέση με άλλε πιο απονευρωμένη, να συρρυκνωθεί κλπ. Εκεί που έχουν ανάγκη αναπτυξιακή κάποια μέρη στην Ευρώπη. Ehm, Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι νέε πολιτικέ. θεωρητικά τουλάχιστον, θα πρέπει να πρικοδοτούνται με νέα κονδύλια. Και οι πρακτικέ πολιτικές όπως η πολιτική συνοχή και όπως η αγροτική πολιτική δεν μπορεί να θεωρούνται απλώς ως ένα λεφτό δέντρο. Όμως τώρα αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συρρυκνωθεί ο προπολογισμό. Επίσης, ταυτόχρονα έχουμε ένα σωρό νέες προτεραιότητες, ένα σωρό νέες ανάγκες. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στον κατάλογο. Οπότε όπως είπα και στην πρώτη ερώτηση, σας ξαναλέω. Οι συνομοθέτες κρατούν το πιδάλιο του προπολογισμού. Αν έχουμε κάποια αλλαγή θετική στο πολιτές πλαίσιο, αυτό θα είναι θετικό και προσωπικά δεσμεύομαι ότι στο σώμα των επιτρόπων θα κάνω ό,τι πρέπει από το χέρι μου. Θα δώσω μάχη ούτω ώστε να κάνουμε αυτό που λέμε. Θα πρέπει όμως όλοι μας να το σκεφτούμε καλά και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Να, σκεφτούμε, να δούμε τι γίνεται με τους ιδίους πόρους, ο Μαρζή. Ευχαριστώ. φίτο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω στην Επίτροπο πως ε, εκτιμώ ιδιαίτερως αυτά τα οποία είπε στην εισαγωγή της ε, γιατί πολλά από αυτά τα οποία είπα ακούγονται ως ε, ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Το ερώτημά μου αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε το θέμα αυτό όσον αφορά τις κοινέ διατάξεις στην ε, πολιτική συνοχή. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια είναι η θέση σας επί του θέματος, ειδικά αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αναλάβει άλλες ε, τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Και δεύτερον, πάντα σε σχέση με την αιρεσιμότητα, η αποχωρούσα κομισιόν πρότεινε μια νέα αίρεσιμότητα αυτή η οποία θα αφορά το κράτος δικαίου που θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διακόψει τα κονδύλια στις ε, χώρες που παραβιάζουν κάποιους όρους. Βεβαίως ε, το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι κάτι τέτοιο δίνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο διακριτικής ευχέρειας και είναι υπερβολικό. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας από αυτού. Σε ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας για την οικονομική σκοπιά. Ως βουλευτής είχα και εγώ την ε, δυνατότητα να επισημάνω τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν αν κάτι τέτοιο ε, ήταν ε, κύκλικο σε σχέση με τον ε, κύκλο της οικονομίας. Ε, τα αποτελέσματα θα τα ένιωθαν ε, δήμοι και περιφέρειες που δεν είναι σε θέση και δεν καθορίζουν την γενικότερη δημοσιονομική πολιτική ενός κράτους. Χαίρομαι λοιπόν και νομίζω πως η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες καλές προτάσεις, αλλά δεν έχει αφαιρέσει το συγκεκριμένο θέμα της μακροοικονομικής ρεσιμότητας. Ε, το σημαντικό είναι να μην υπάρχει κάποιος αυτοματισμός και για την αιρεσιμότητα του κράτους ε, δικαίου. Θα πρέπει να θυμάμαστε την αρχή της αναλογικότητας. Οπότε ε, δεν θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει κάποιος αυτοματισμός. Είναι ευαίσθητο το θέμα, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Και υπάρχει και μια άλλη πτυχή ευαίσθητη. Αν υπάρχει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, η Κομισιόν μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο να ανασταλούν ε, οι πληρωμές ή να σταματήσει η ανασταλή των ε, πληρωμών. Βεβαίω εμείς μιλάμε ε, πάντα με βάση τους κανόνες και το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Η διαχείριση δε των κονδυλίων αυτών απαιτεί ότι οι χώρες ε, θα πληρούν ε, τους βασικούς ε, κανόνες μιας δημοκρατικής λειτουργίας. Να υπάρχει κίνδυνος μια χώρα να μην ανταποκρίνεται σε αυτά, τότε είναι ευθύνη της Κομισιόν να ερευνήσει και πιθανώς να αναστείλει τις πληρωμές. Αυτά είναι τα δύο θέματα που θίξετε, αυτή την απάντηση μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σχετίζεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Εθνική Συγχρηματοδότηση. Εσείς ε, λέτε πως ε, θα ήταν χρήσιμο να ε, συζητήσουμε το πώς θα μπορούσαν να αποκλειστούν από το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, οι εθνικές ε, συγχρηματοδοτήσεις ε, του Ταμείου Συνοχής. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η εντολή την οποία λάβαμε από την επιλεγήσα ως πρόεδρο είναι να υπάρξει μια ευελιξία στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητάτε είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, υπάρχει ένας ε, χρυσός κανόνας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένες προτάσεις, γιατί ούτως ή άλλως το ζήτημα αξιολογείται εντός Κομισιόν και θα παίξω και εγώ ενεργό ρόλο μαζί με τους ε, συναδέλφους μου για το πώς θα συνεργαστούμε με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τον ε, υποψήφιο επίτροπο για την οικονομία. Πρέπει να δούμε το σύμφωνο. Δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να απορρίψουμε ή να δεχτούμε κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το δούμε συνολικά. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων με την Μαρτίνα Μίχελς για την Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά και Βορεια Πράσινη Αριστερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φερέρα. Οπωσδήποτε χαίρομαι για την φιλοδοξία που επιδεικνύεται και πάλι και σήμερα μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία στο νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχής αλλά λυπούμε λίγο για το ότι στις γραπτές σας απαντήσεις δεν ασκείται καμία κριτική και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις προτάσεις της προηγούμενης ε, Κομισιόν. Αφενός ε, δηλαδή τον ε, περιορισμό σε δύο προτεραιότητες, σε καινοτόμο οικονομία και ψηφιοποιημένη και την προστασία του κλίματος. Ε, τι βλέπετε εσείς όμως να γίνεται στην πλευρά της κοινωνικής συνοχής, ε, του οικολογικού και κοινωνικού ε, μετασχηματισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Κύρια Βουλευτά, δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα την ερώτησή σας, αν αναφέρεστε στην σύνταξη της πρότασης της Κομισιόν, γιατί αυτά που είπατε καλύπτονται. Υπάρχει σαφής αντίληψη του ότι όταν παρεμβαίνουμε κάπου πρέπει να συνδυάσουμε τα κοινωνικά στοιχεία με τα κλιματικά και τα οικονομικά. Αυτό είναι ο συνδυασμός που θα κάνει την σύγκληση αποτελεσματική. Αλλά αν δεν ε, σας κατάλαβα, σας παρακαλώ να διευκρινίσετε. Κοιτάξτε, εγώ αναφέρομαι στον στόχο που περιέχει η συνθήκη της κοινωνικής συνοχής και της σύγκλησης των συνθήκων ζωής, ε, η οποία θεωρώ ότι παραλείπεται εδώ πέρα από τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, γιατί ως Ευρωβουλευτής ε, δικαίως ε, τότε αναδείξατε το πρόβλημα αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Μπορείτε να μας περιγράψετε συγκεκριμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν θα μετράνε μόνο τα πλεονάσματα αλλά και το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια σύγκληση και μια βελτίωση των συνθήκων ζωής. Σας ευχαριστώ. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, για εμένα, το πλαίσιο αυτό, είναι ένα μέσο για να επιτρέψουν στις χώρες ε, της ε, Ευρωζώνης και τις χώρες που θέλουν να μπουν στο ευρώ να είναι σε οικονομική θέση να κάνουν τα ουσιαστικά για την ε, σύγκληση. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, δεν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις που θα επιβάλλονται. Νομίζω πως το είπα σαφώς ότι πρέπει οι προτάσεις να συζητούνται με το Κοινοβούλιο. Αλλά όταν κάποιο είναι σε ένα κοινό και υπάρχει μια προσαρμογή και είναι δύσκολο για τις χώρες να ανταποκριθούν στις απαιτήσει για τα υγιή, δημόσια, οικονομικά, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα μπορούν γρήγορα να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαμε κάποιες θετικές εμπειρίες. Ε, τεχνική στήριξη που δόθηκε σε διάφορες ε, χώρες, ε, η κατάρτιση, μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης του φορολογικού συστήματος. Όλα αυτά είναι διαφορετικές πτυχές και θα είναι ακριβώς η ίδια μονάδα η οποία θα ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Να τα πω αγγλικά. Έχουμε τις, ε, τα προγράμματα, τα εθνικά μεταρρυθμίσεων ε, ή τα προγράμματα ε, που αφορούν τις συστάσεις χώρα Στο παράρτημα Β έχουν πολύ περισσότερα πράγματα πλέον από ό,τι είχαν στο παρελθόν, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα για να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία. Και εδώ πέρα απαιτείται η εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Όλοι θα πρέπει να εμπλακούμε πολύ περισσότερο να δούμε προληπτικά όσον αφορά το τι θα περιέχουν αυτές οι συστάσεις και να ταιριάζουν βεβαίως στην κάθε χώρα. Μιλάμε για την διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε μια ατζέντα σοβαρή για να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω χωρών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να πηγαίνουν και να συνδυάζονται με τις αρχές της συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Θα αφήσω ε, καταρχάς ε, τον κύριο Πασκάλα Ριμό να κάνει την ερώτησή του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, ε, κυρία Φερέρα, Ε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από το να του χωρίς στα πορτογαλικά και θα συνεχίσω στα γερμανικά. Σε ό,τι αφορά τη διασυνορική συνεργασία, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πολύ καλά το πρόγραμμα Interreg, το οποίο θέλει να ε, δημιουργεί γέφυρες φιλίας και όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών. Το Ιντερεκ βοηθά όχι μόνο να ε, φαίνονται λιγότερο, γίνονται λιγότερο αισθητά τα φυσικά σύνορα, αλλά να μην είναι και τόσο αόριστη για τους πολίτες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόνα. Λυπούμε την προβλέπερη κοπή αυτών των κονδυλίων για την επόμενη περίοδο κατά 30% από 10,2 σε 7,6 ε, Και μετά το 2020, αν λέει ε, αυτό που λέει γραπτή σας απάτη, δεν με βρίσκει σύμφωνος ότι θα ήταν κάτι ε, επαρκές. Ε, όχι. Αν τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο και μεγαλύτερο εθνικισμό, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα για την υπερκέραση των συνόρων. Και μια ερώτηση, θα είστε στο πλευρό μας ώστε τουλάχιστον ε, να διατηρηθεί ε, η πρικοδότηση στο επίπεδο του Συμβουλίου και δεύτερον ε, σε ό,τι αφορά αυτές τις διαπεριφερειακές καινοτόμες επενδύσεις. Σας φαίνεται καλή αυτή η ιδέα για τα Component 5 που θα πάνε στο άλλο ταμείο και για το Interreg Europe Το έχει διαγράψει εντελώ ε, η Κομισιόν αυτό το πρόγραμμα. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ στα γερμανικά μόνο ευχαριστώ μπορώ να σας πω. Πάω στα πορτογαλικά λοιπόν για την απάντησή μου και θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση σε αυτά που είπατε. Γιατί είπατε ότι στη γραπτή μου απάντηση Λέω ότι είναι επαρκή η είναι ενδεδειγμένη μείωση. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι η πρόταση αυτή είναι ενδεδειγμένη, αλλά ληφθούν υπόψη διάφοροι περιορισμοί. Δεν είπα ότι μ' αρέσει που υπάρχει αυτό ο περιορισμό, αλλά είπα ότι η πρόταση αυτή ε, είναι με επαρκή πρόταση για να μπορέσουμε πάνω σε αυτή να δουλέψουμε. Αυτό ήθελα να πω και επαναλαμβάνω κάτι που είπα και πριν. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που θα πρέπει να ορίσει φιλόδοξου ε, στόχου ε, και τιμέ, και έπειτα αυτοί να μειώνονται. Να μειώνονται τα κονδύλια και τελικά να καθυστερούν και οι εργασίες για το ΠΔΠ. Λοιπόν, έρχομαι στο Interreg που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίς καμιά αμφιβολία πρόγραμμα το 1990 κάτι είχα εργαστεί στο πρώτο πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας με τη Γαλλικία, την ισπανική αυτή περιφέρεια και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία δεν ε, θεωρώ ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μειώσει ε, το ίντερεκ. Το αντίθετο, νομίζω ότι θα συνδυαστούν τα κονδύλια του προπολογισμού για να μπορέσει να παραμείνει το ίντερεκ έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε διατεθειμένοι προ αυτό. Δεν μπορώ βέβαια να σα πω κονδύλιο προ κονδύλιο του προπολογισμού ακριβώ τι θα γίνει. Δεν ε, ξέρω ακριβώ τι γίνεται με την ευελιξία. Πάντω, ε, αυτό που θέλουμε, μπορώ να σα το πω, είναι να δώσουμε, ε, να ενισχύσουμε περισσότερε πρωτοβουλίε δυνάμει του Ιντερνετ. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό. Θέλουμε να καταρρύψουμε τα πολιτικά σύνορα που υπήρχαν. Θέλουμε να μπορούν να συμβιώνουν οι γείτονε ε, από τη μια χώρα στην άλλη. Και το ίντερνετ γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό ο του. Δεύτερη ερώτηση. Ε, θα ήθελα την άποψή σας για ένα θέμα της επικαιρότητα, φυσικά το Brexit. Ε, το Interreg μεταξύ άλλων ε, χρησιμοποιείται από το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν 500 προγράμματα του Ιντερεγ. Αν υπάρξει αυτή η αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, και επειδή συμμετέχει η ε, Βόρειος ε, σε πολλά από αυτά τα προγράμματα, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα το τι θα γίνει και ιδίω σε περίπτωση άτακτου Brexit ε, με τις υποχρεώσεις της Μεγάλης Βερτανής για αυτά τα προγράμματα. Ε, τα πράγματα με τα σύνορα είναι προβληματικά, υπάρχει ένα πρόβλημα και καλό είναι να υπάρξει συνεννόηση για την επίλυση λύσεων. Θα πρέπει να υπάρξει κοινή οργάνωση, θα πρέπει να υπάρξει συνομιλία και συνδιαλλαγή αλλαγή. Οι σχέσεις, τα προγράμματα ε, μπορούν να κινδυνεύσουν και αν ε, έχουμε ένα σκληρό Brexit, έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο κομισιών. Απάντηση. Όπως τα γνωρίζετε, δύσκολο το σχέδιο από τώρα για το Brexit χωρίς συμφωνία, περίπλοκο το θέμα, ούτε ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες από τέτοιο Brexit. Το Ταμείο Αλληλεγγύης θα ενεργοποιηθεί υπό ορισμένους όρους. Όμως θα πρέπει να υπάρξει κατεπίξω βοήθεια σε κάποιες ε, περιοχές, σε κάποιες περιφέρειες, σε κάποιες χώρες που θίγονται. Και έτσι να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε τις αρνητικές συνέπειες από ένα τέτοιο ε, Brexit χωρίς συμφωνία από το ε, αδιαπέραστο σύνορο. Ε, όχι βέβαια, είναι ανεπιθύμητο και αν γίνει τότε θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε όλα, όλα υπό το Interreg και ό,τι οτιδήποτε συμφωνία συνεργασίας υπάρχει. Να δούμε υπάρχουν αρκετοί πόροι για να έχουμε τελείω ε, καινούριο το ελληνικό σύστημα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για τι ε, πλησόμενε εταιρείε. Εδώ μέχρι και προσωπικές σχέσεις πρόκειται αυτό το αδιαπέραστο σύνορο να χτύπηθουν. Τόσα ξέρω, τόσα σας λέω, αλλά δεν νομίζω ότι κανένα ξέρει ε, πού θα οδηγηθεί η κατάσταση και υπό ποιου όρου θα γίνουν όλα αυτά. Το παρακολουθούμε από κοντά. Και τώρα. Ιζαμπέλ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Καρβαλιά, είπε η Επίτροπο, είπατε τέλο πάντων κύριε Επίτροπε, ότι θα συνεχίσετε τις βασικές πολιτικές, τη σύγκληση, τη συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, επενδύσεις, αλλά θα πράγματι τι γίνεται και με τις ε, διαδοτικές μεταρρυθμίσεις που πάντοτε πρέπει να συνοδεύονται από επενδύσει. Πώ αυτά θα τα συγκεράσετε. Γιατί υπάρχουν και πράγματα αλληλοσυγκρόμενα. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων θα οδηγεί σε περισσότερη συνοχή θέση εργασίας, καλύτερες δεξιότητες για τον κόσμο, καινοτομία και ταυτόχρονα να μην έχουμε οικονομία άνθρωπη. Ευχαριστώ βουλευτά, λέει η Επίτροπος. Επί Μακρόν συζητούμε και επιδιώκουμε οικονομική θωράκιση της Ευρωζώνης. Το κοινωνόμισμα οδήγησε σε ανοιχτούς ανταγωνισμούς. Χωρίς να υπάρχουν περιθώρια για αντίμετρα ούτως όπως υποβάθμιση και άλλα σταθεροποιητικά μέτρα, οπότε ε, χωρίς να υπάρχει τέτοιο σύστημα θα είχαμε οδηγηθεί σε μεγαλύτερη κρίση. Επίσης ε, έχουμε και κάποιες ανισορροπίες μεγάλες μεταξύ κρατών μελών, οπότε θέλουμε αυθεντική σύγκληση. Όμως χρειάζονται πετυχημένες πολιτικές επενδύσεις και έτσι να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να κινηθούν προς την σωστή κατεύθυνση ταχύτερα. Και όταν μιλάμε για διορθωτικές μεταρρυθμίσεις, τότε μιλούμε για μεταρρυθμίσεις που είναι δυνατόν και πρέπει να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και θα πρέπει κατά να τις εξετάσουν και να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται και όλοι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι να ξέρουν τι προτείνεται, να υπάρχει κάτι σαν συμβόλαιο με αυτές τις χώρες. Αν πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, θα αμείβονται. Είμαι επικεφαλής δύο γενικών διευθύνσεων για συνοχή και για μεταρρυθμίσεις. Και αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις σε κάθε περιοχή. Οι δύο πτυχές αυτού του θέματος δεν θα πρέπει να αντιφάσκουν. Θα πρέπει μάλλον η μία να υποστηρίζει την άλλη. Είναι και θέμα δημοσία διοίκηση και έτσι θα πάμε σε μια πετυχημένη πολιτική συνοχή και σε μεγαλύτερη συνοχή. Βέβαια και το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να βοηθήσει. Θα έχουμε καλύτερους ανθρώπινους πόρους και αυτό θα βοηθήσει συνοχή. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσύνθεση ε, και όχι αντιφατικότητα μεταξύ των δύο αυτών ε, πολιτικών. Σε όλα αυτά θεωρητικά βοηθάει το ενίο νόμισμα, το λέει και η συνθήκη, συνοχή έχουμε, προβλέπεται, αλλά θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε για το ευρωπαϊκό όραμα. Και, λέει κυρία Καρβαλιά, σε επερώτηση, όμως, όμως, πώς θα χρησιμοποιήσετε το εξάμεινο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Για πέστε μας δύο λόγια. Να μην ξεχνούμε τι προβλέπει το εξάμεινο τι λένε οι συστάσεις για κάθε χώρα. Επιταχύνεται έτσι η σύγκληση. Και να μην ξεχνούμε ότι όταν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις υλοποιούμε δεν θα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη με κάθε κόστος. Θα πρέπει να δούμε ότι πρώτα πρώτα έχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης πάνω απ' όλα, η ισορροπία. Δεν είναι δυνατόν να σκεπτόμαστε μόνο τα ποσά και τα, τους αριθμούς και όχι την ποιότητα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Επόμενος. Πρόεδρος Κριστιαν Κινέα. Ε, despite all the talking about simplification, both Τα όσα ακούγονται για την απλοποίηση και εδώ στις Βρυξέλλες και στα κράτη-μέλη οι δικαιούχοι εξακολουθούν να παραπονιούνται για υπερβολική γραφειοκρατία. Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι δικαιούχοι θα δουν πραγματική απλοποίηση επιτόπου. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφέρατε στην αρχική σας ε, τοποθέτηση το ε, απλοποιημένο ε, κόστος. Για να είμαι ειλικρινής, με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Ήμουν και υπουργό στη Ρουμανία όταν ξεκίνησε, αλλά είναι και ένα πρόβλημα γιατί ε, υπονομεύθηκε η λύση από τις πιθανές μελλοντικέ αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που γνωρίζω ότι είναι ανεξάρτητο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει και μια σταθερότητα για τους δικαιούχους. Ε, θα συνεργαστείτε με το ελεγκτικό συνέδριο για να μην μπλέξουν σε διαφορετικές ερμηνείες οι δικαιούχοι. Σας ε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, αυτό το οποίο με ρωτάτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιος μου είπε άτυπα πως ε, οι μικρές ε, εταιρείες πλέον δεν ασχολούνται με την κοινωτική στήριξη γιατί δεν μπορούν δεν έχουν το προσωπικό για να ασχολείται με όλη την ε, γραφειοκρατία. Αυτό είναι αντίστοιχο με τους στόχους ε, που έχουμε θέσει. Έτσι. Ακριβώς το σκεπτικό μας είναι η πολιτική μας να φτάνει στους ανθρώπους ε, επιτόπου. Τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν πρέπει να προσαρμοστούν εάν δεν επιτυχάνουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Πιθανώς θα έρθουμε σε επαφή με τους δικαιούχους να τους ρωτήσουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να απλοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τους όρους ε, πιο εύκολους ε, στο να τους εκπληρώνετε. Δηλαδή να το δούμε από τη σκοπιά του πελάτη ε, τρόπον τι ε, να δούμε και ποιες από τις απαιτήσει αυτές είναι αγκαίες και ποιες όχι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε όμως να εξασθενήσουμε τις δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι τα λεφτά ξοδεύονται σωστά. Υπάρχουν απαιτήσει ε, νομικές ε, της συνθήκης ε, για το πώς θα πρέπει να ξοδεύονται τα λεφτά έτσι. Δεν δηλαδή, μιλάμε για απλοποίηση, αλλά υπάρχει και αυτό. Σας ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τις δύο ιδιότητές σας, γιατί θα έχετε ε, ένα χαρτοφυλάκιο που λέγεται συνοχή και μεταρρυθμίσεις και υπάρχει και μια νέα γενική διεύθυνση στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, για να είμαστε πιο σαφείς, κάποιοι λένε ότι θα υπάρχει μια de facto αιρεσιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται μεταρρυθμίσεις για να εκταμιευτούν κονδύλια συνοχής. Ε, ισχύει αυτό ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι φωνές αυτές ε, μεταφέρουν έναν φόβο ότι θα υπάρξει μια επιπλέον αιρεσιμότητα στα ταμεία και ότι τα ταμεία θα υπαχθούν στις μεταρρυθμίσεις. Θα προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι πρώτα απ' όλα οι μεταρρυθμίσεις θα είναι επαρκείς και θα θεωρούνται αναγκαίες από τα κράτη-μέλη, ότι τα κράτη-μέλη θα αντιλαμβάνονται πλέον θα προτείνουν μεταρρυθμίσεις και ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ε, θα συνεισφέρουν σε μια αύξηση της δυνατότητάς τους να αναπτυχθούν ε, και στην αύξηση της ταχύτητας σύγκλησης. Άνα δούμε προσεκτικά τη δουλειά που έχει γίνει στο πλαίσιο αυτού του μεταρρυθμιστικού πακέτου στο παρελθόν και το αναφέρω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό. Η δουλειά η οποία γινόταν από αυτή την μονάδα ε, υποστήριζε πάρα πολύ την Ελλάδα, τη Λιθουανία και θεωρείται το πολύ θετική και μπορώ να σας πω ότι ε, λειτουργούσαν ε, μόνο στην τεχνική στήριξη 26 χώρες ε, και είχαν προτάσεις που διπλασίασαν τις ε, ικανότητες ε, των μονάδων για τεχνική στήριξη. Οπότε είναι... έχουν μια πάρα πολύ θετική εικόνα. Λοιπόν, θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η στήριξη, αλλά υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο, η δυνατότητα επενδύσεων. Λοιπόν, θεωρώ ότι λύνουμε ένα πρόβλημα και δημιουργούμε ένα νέο μηχανισμό που θα βοηθήσει την νομισματική ένωση να λειτουργήσει με λιγότερους ε, κινδύνους ε, από ό,τι μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο εξαιρετικέ ερωτήσει. Το λόγο τώρα έχει ο συνάδελφος Άλβαρο Αμάρο. Ευχαριστώ. Senhora Comissária do Estado, cumprimento, cumprimento Presidente e todos. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια κύριε Φερέρα. Εγώ θέλω να πω το εξή. Ήρθα σε αυτήν την ακρόαση με έκπληξη από όσα είχα διαβάσει και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί μου προξένησαν ανησυχία ορισμένα από αυτά που διάβασα. Πρώτα απ' όλα, ως Ευρωπαίος πολίτης, ε, αν εσείς ε, έχετε την πολιτική βούληση και την πολιτική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχετε, υποθέτω, θα έπρεπε να έχετε και τη σιδηρά βούληση να αποφύγετε αδικίες. να δεχθείτε να βοηθηθούν οι πιο πλούσιες χώρες σε βάρος των πλέον αδύναμων και φτωχών ε, είναι άδικο. Εγώ ως Πορτογάλος τα βλέπω και από τη δική μου την οπτική γωνία τα πράγματα. Με εξέπληξαν αυτά που διάβασα. Βέβαια, ακούγοντάς σας διασκεδάστηκαν οι ανησυχίες μου και έρχομαι στο ερώτημά μου. Μπορείτε να υπογράψετε τη δέσμευση αυτή με τις πιο φτωχές περιφέρειες. Απάντηση, μην ανησυχείτε. Καθόλου μην ανησυχείτε. Διότι δεν είναι κάτι καινούριο η προσήλωσή μου στα θέματα της συνοχής. Του, του, του λεχθέντος αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν θα επεξεργαστούμε την πρόταση της Κομισιόν όπως την παρουσίαση ή αν θέλουμε μια άλλη πρόταση. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα έγγραφο εργασίας. Χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει όμως με τα έσοδα του υπολογισμού. Δηλαδή το έγγραφο αυτό έχει συνταχθεί με βάση μια λογική υπόθεση, μια εύλογη υπόθεση. Και ξέρουμε ότι θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες από τις χώρες που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρόβλημα της αποχώρησης ενός ε, καθαρού συνεισφέροντος. Και αυτό θα δημιουργήσει τρύπες στον προϋπολογισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης έχουν τον λόγο των συνόρων, την ασφάλεια, την άμυνα, την πολιτική γειτονία, ε, Ευρώπη στον κόσμο. Είναι και αυτά προτεραιότητες. Εγώ σε εσά έχω στρωμένο το βλέμμα μου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στο Συμβούλιο βέβαια και στο πώς θα τα βρείτε μεταξύ σας. Και φυσικά θα αγωνιστώ ώστε το Συμβούλιο στις επαφές που θα έχει με το Κοινοβούλιο και στις ε, διαβουλεύσεις και ξέρω ότι πολλοί από εσάς εργάζεστε για χρόνια σε αυτά τα θέματα, θα φροντίσω λοιπόν να βοηθήσω ώστε να βρεθεί λύση στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα και προσήλωση. E ναι, έχετε εσείς στραμμένο το βλέμμα ε, σε εμά, αλλά εμείς έχουμε στραμμένο το βλέμμα σε εσά. Διότι αν η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μας μιλάει για λιγότερο πικροκατοικημένες περιφέρειες, γιατί μιλάει τελικά. Δεν μιλάει για τη συνοχή. Τι προσδοκίες υπάρχουν. Εσείς αν αναλάβετε τη θέση αυτή στην Επιτροπή, ε, πιστεύω ότι όταν μας λέτε τι πιστεύετε, ε, τα εννοείτε και σας πιστεύω. Το πρόβλημα είναι οι δυσκολίες που είναι πραγματικές. Τι θα γίνει. Η πολιτική συνοχή ε, κατοχυρώνεται στις συνθήκες. Πράγματι μπορεί να υπάρξουν τρύπε στα έσοδα, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει τρύπα στην πολιτική συνοχή, γιατί αυτό θα σημάνει μεγαλύτερη αδικία στην Ευρώπη. Άρα, αυτή την αποφασιστικότητά σας, την προσήλωσή σας, πρέπει να τον αξιοποιήσετε για να μην μειωθούν τα ποσοστά χρηματοδότηση ούτε για τι λιγότερο κατοικημένε περιοχέ. Απάντηση, ακούστε. Του πόρου δεν του ορίζει η Κομισιόν, αλλά το Συμβούλιο. Άρα αυτούς πρέπει να πείσουμε και τα κράτη-μέλη, γιατί αυτοί πρέπει να συνεισφέρουν στον προπολογισμό. Πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο στον προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα συμμετοχής, και συγχρηματοδότησης, ε, ξέρετε ότι αυξήθηκαν για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης το 2009. Τώρα θα πρέπει να δούμε, γιατί σιγά σιγά επανέρχεται η ομαλότητα. Και έχουμε το χρονοδιάγραμμα, έχουμε το πρόγραμμα προσαρμογής, αν θέλετε, για να μην υπάρξουν ε, προβλήματα.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 Αγαπητή κυρία Φερέιρα, ως ε, μία από τις ε, νέες ερχόμενες εντός αγωγικών χώρες της Ένωσης, η Βουλγαρία, όπως και πολλές άλλες χώρες, ε, ωφελήθηκε τα μάλα από την πολιτική συνοχή. Ωστόσο, η Βεροδυτική Βουλγαρία είναι από τις φτωχότερες ε, περιφέρειες της Ένωσης Πιστεύω λοιπόν ότι οι πολιτικέ πολιτικές θα μπορούσαν, μάλλον οι ενωσιακέ πολιτικέ μπορούσαν να συνδυαστούν και να συμπληρώσουν τις εθνικές προσπάθειες, αντιμετωπίζοντα οικονομικέ ε, δημοσιονομικέ και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένε περιφέρειες. Τι μέτρα λοιπόν θα μπορούσατε να, να εφαρμόσετε για να στηρίξετε τις χώρες κεντρική και ανατολική Ευρώπης ε, για να φτάσουν στο μέσο επίπεδο διαβίωση τη Ένωση. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω απάντηση ακριβώς σε αυτά τα προβλήματα είναι πολιτική συνοχή. Εγώ βέβαια δεν θέλω να πω με αυτό ότι θα είναι κάτι πολύ ε, εύκολο και γρήγορη αλλαγή οικονομικής ε, <clears throat> διάρθρωσης ε, των περιοχών που υπολείπονται και σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες ε, και σε ό,τι αφορά τη διάθεση των παρκών κονδυλίων. Η πολιτικές συνοχής όμως πρέπει να εστιάσει αυτές τις περιφέρειες που υστερούν, που υπολείπονται και θα πρέπει να εργαστούμε σε συντονισμό και με άλλες πολιτικές. Δεν μπορεί η πολιτική συνοχής να είναι απομονωμένη από την κοινωνική πολιτική, από την οικονομική πολιτική. Και θα πρέπει όταν ξέρουμε τις λεπτομέρειες για μια περιφέρεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγει από την κατάσταση αυτή. Παραδείγματος αν χρειάζεται βοήθεια για την επαγγελματική κατάρτιση μια περιφέρεια ή μπορεί να χρειάζεται θεσμική ενίσχυση ή ανανέωση των υποδομών ή οτιδήποτε. Άρα η πολιτική συνοχή θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις περιφέρειες και στις ανάγκες τους. Και θα πρέπει να εστιάζει ακριβώς στο τοπικό επίπεδο και να αναζητεί τα πλέον κατάλληλα μέσα παρέμβασης. Νομίζω αυτό είναι μια εξαιρετική βάση εργασίας. Και είναι σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, διότι πολλές από τις χώρες μας ε, έχουν βιώσει ή βιώνουν ακόμη τέτοιου είδους εμπειρίες. Γι' αυτό λοιπόν διαπεριφερειακή συνεργασία είναι θεμελιώδης, για να μπορέσουμε ένας να διδαχθούμε από τον άλλο και να μην παραλάβουμε λάθη, σφάλματα του παρελθόντος. Αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να μας διέπει. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω, αυτή είναι η αρχή μας. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο οι περιφέρειες θα μπορέσουν να φτάσουν σε μια ε, ταχύτερη σύγκληση για να προσεγγίσουν αυτές που βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο. Δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, που έχει να κάνει με τις γραπτές σας απαντήσω, που λέτε ότι συμφωνείτε με την προτινόμενη περικοπή της τάξης του 10% για την μακροχρόνια πολιτική συνοχής. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα η πρόταση για αύξηση των εθνικών ποσοστών συγχρηματοδότησης. Πώς αυτά τα μέτρα θα επηρεάζουν τις που έχουν οι πιο φτωχές περιοχές της Ένωσης να ζητήσουν και να λάβουν υποστήριξη για να έχουν πιο ταχύ οικονομική ανάπτυξη. Απάντηση. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα ήδη. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν βασίστηκε σε μια μεγάλη μείωση αυτή ήταν υπόθεση εργασία, δηλαδή. Αυτό το νέο ποσοστό συγχρηματοδότηση είναι κάτι καινούριο πράγματι. Αυξήθηκαν τα ποσοστά αυτά, διότι σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης τα κράτη-μέλη δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν την εθνική χρηματοδότηση και οι εργολάβοι δεν μπορούσαν να εφαρμόζουν τα έργα τα οποία έπρεπε να υλοποιηθούν. Ήταν πολύ περιορισμένες ε, οι δυνατότητες. Τα κρατικά ταμεία δυσκολεύονταν και εξακολουθούν κάποιες χώρες να μην έχουν περιθώρια λιγμών. Αλλά σταδιακά αυτό που θέλουμε είναι να εξομαλύνουμε την κατάσταση με τα ποσοστά συγχρηματοδότηση, εφόσον ανακάμπτει από τη φαίνεται η οικονομία, επανέχεται στην ομαλότητα όπως είπα. και στην κανονικότητα. Μπορεί η μόχλευση τώρα να βοηθήσει Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά είναι καλά σε αυτή την πρόσβαση στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και νομίζω χρηματοδότηση καλά, σε καλ, με καλού συντελεστέ. Είναι κάτι καλό που μπορεί να βοηθήσει του ε, εργολάβου. Καρολίν Ροζ. Καρολίν Ροζ. Κυρία υποψηφία επίτροπε, τα τελευταία χρόνια διαπιστώσαμε ότι έχει χρηματοδοτήσει η Ένωση ένα σωρό προγράμματα για το περιβάλλον, και αυτό κόντρα στις απόψεις των ντόπιων πολλές φορές προτιμήθηκαν οικονομικά συμφέροντα και όχι το περιβάλλον ή η κοινωνία κράτη-μέλη ε, επιδοτούν ε, ορυκτά καύσιμα που χειροτερεύει την κατάσταση για το κλίμα. Τι γίνεται στα πλαίσια της κρίσης για το κλίμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα πρόγραμμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και προτείνουμε στα πλαίσια της Digi Region υπάρχει μια υπηρεσία η οποία να είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον, στα οικονομικά συμφέροντα και να βρίσκει την λύση στις συγκρούσεις μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Τι γίνεται με τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Πώς το βλέπετε, δεν πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ταμείο για να, χρησιμο... να, να χρηματοδοτούμε κάποιους αυτοκινητοδρόμους που υπάρχει και στο Στρούμα, στην... Ε, στο Στριμώνα στη Βουλγαρία, τέλος πάντων, που υπάρχει αυτοκινητόδρομος, αλλά είναι ζώνη προστατευμένη περιβαλλοντικά. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και... Βεβαίως, βεβαίως. Θα το κοιτάξω και θα σας πω, όπως φαντάζεστε, ότι θα κάνω. Και δεν έχω πιστεί ότι έχουμε επενδύσεις σε προγράμματα που βλάπτουν το περιβάλλον. Απλώς, όπως με τα ανθρακοριχεία, δεν έχουμε πια λεφτά για τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ή κάποιο αεροδρόμια. Τόσο αεροδρόμια είναι στην απότερη περιφέρεια. Οπότε, οπότε έτσι γίνεται. Και μας είπατε για κάποιον αυτοκινητόδρομο, και στο Στριμώνα, Στρούμα. Θα πρέπει να το δω και να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Είναι σημαντικό η κοινωτική νομοθεσία να τηρείται. Θα πρέπει δε να έχουμε τα προγράμματα που χρειάζονται πάντοτε όμως να διαπνέονται από τις αξίες μας. αν προστατεύεται ε, από την UNESCO ή από οποιοδήποτε πλαίσιο μια περιοχή, φυσικά και πρέπει εμεί να συμμορφωνόμαστε και όταν χρειάζεται να βρίσκουμε εναλλακτικέ. Ό,τι είναι λιγότερο βλαπτικό. Να λαμβάνουμε μέτρα που να περιορίζουν το κακό, όποτε υπάρχουν απόφεκτες ε, συνέπειε. Οπότε βέβαια το πρώτο είναι να τηρείται ο νόμος. Αλλά θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε κάθε πρόγραμμα χωριστά και να μην υπάρχει ανισορροπία να γίνεται ένα καλό και ένα κακό, ας πούμε, τη βάρος του περιβάλλοντος. Αλλά θα πρέπει πρώτα να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Θα πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, προσβασιμότητα. Οπότε δεν μπορώ τώρα στο γόνατο να σας πω την απάντηση, αλλά θα το δουν οι συνεργάτες μου και θα σας πούμε Ευχαριστούμε. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να έχουμε καλύτερους μηχανισμούς για τη συμμετοχή και την βιωσιμότητα. η τρική σχέση. Από τι πνεύμα διαπνέεται. Νομίζετε ότι όλοι οι ενεχόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία των ιδιωτικών ταμείων. Δηλαδή το 20 θα είναι κρίσιμη καμπή για την συμμετοχή των διαφορών εταίρων και η χρηματοδότηση θα σχεδιαστεί από τα κρατημέλη, αλλά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέει για εμπλοκή των ντόπιων, αλλά αυτό προποθέτει κάποιους μήνες. Άρα πώς θα γίνει εταιρική σχέση. Θα μείνουν απ' έξω οι ενεχόμενοι οι εμπλεκόμενοι και οι θυγόμενοι. Άρα θα πρέπει όλους να τους λάβετε υπόψη. Όλα αυτά θα πρέπει να λάβετε υπόψη για το πρόγραμμα του 2020. Τι γίνεται με τον κώδικα διοντολογίας. Απλώς νομικής, τι ισχύει, τι θα γίνει το 2020. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι η εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική. Ναι. Να υπάρχει συνεργασία με τους ντόπιου. Θα το ψάξω. Θα δω τι ισχύει. Από ό,τι ξέρω, όντως οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει να εμπλέκονται ούτως ώστε να υλοποιούνται τα προγράμματα και αυτό είναι καλό για όλους. να συμμετέχουν οι τοπικοί πλήρως σε όλα τα προγράμματα. Εγώ έχω συμμετάσχει και έχω δει να συνεργάζονται τα συνδικάτα, ε, οι φορείς ε, των επιχειρήσεων, η ΜΚΟ, όλα αυτά ήταν προσθεμένη αξία. Όλα αυτά είναι παραγωγή Πάντω για το τι ισχύει τώρα θα το ψάξω και θα δω. Όλα αυτά πάντως είναι πάγιες αρχές που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντρού. Euh, Κύριε Επίτροπε, παρά το στόχο της περιφερειακής συνοχής έχουμε κάποιες ε, περιοχές που παραμένουν φτωχές, Ακόμα δεν έχουμε την καλή διαχείριση των πόρων στην περιφέρεια ή στην απότερη περιφέρεια. Έχουμε μεγάλη φτώχεια και ανεργία. Καμιά φορά εντυπωσιακέ. Να, για παράδειγμα, έχουμε 40% στην ίσο που είναι κάτω από το. Ε, κάτω τη φτώχεια, 24% άνεργοι. Στη Γαλλία είχαμε το Μάιο μια μελέτη που έλεγε ότι η διαχείριση των ταμείων στην Ευρώπη ε, γνώρισε αύξηση του κόστου διαχείρισης και μείωση της ε, αποτελεσματικότητα. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε τόσο ώστε όλοι αυτοί ε, να βοηθηθούν οι άνθρωποι και να πιάνουν τα χρήματα των Ευρωπαίων και τι γίνεται για την απότερη περιφέρεια. Τι, τι νομοθέτημα μπορεί να υπάρχει για να βοηθηθεί η οικονομία τους. Πώς μπορεί οι εισαγωγέ να φορολογηθούν και να τι βοηθήσουμε. Προσοχή με τις ε, επιδόσεις συγγνώμη, με τις επιδοτήσεις ε, και τις εξαιρέσεις που προβλέπουν για αυτές τις περιφέρειες, διότι άλλωστε υπάρχει και το άρθρο 343, το οποίο προβλέπει σχετικά η Επίτροπος οι περιοχές τη απότερης περιφερειάς όντως είναι προτεραιότητα. Ακριβώς, όπως είπατε το άρθρο 343 το ορίζει τούτο. Ορθώς είναι προτεραιότητα και για μας. Το είπε και η νέα πρόεδρος Επιτροπής και μας επέσυρε την προσοχή. Να προσέξουμε ιδιαίτερος. Να προσέξουμε την ανάπτυξη αυτών των ε, τόπων. Είναι μακριά. Δύσκολη πρόσβαση. Είναι εξαιρετική φύσης η κατάσταση. Εντάξει, εξαίρεση και για τα αεροδρόμια προβλέπουμε θέματα ε, επίσης μετρολογικά και έχουμε εκπονήσει 21 προτάσεις. Αυτές αφορούν ακριβώς την αποτελή περιφέρεια από διαφορετικές πλευρές. Ε, προβλέπουμε την ευκολότερη πρόσβασή τους ε, στα κονδύλια. Έχουμε χαμηλά κατόφλια για ενίσχυση του κόσμου, της αλληλείας, και η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει για αυτές τις περιοχές να λάβει υπόψη τη σχέση μεταφορών και περιβάλλοντος, αλλά και άλλων πολιτικών. Πολλές φορές έχουμε μόνο εκεί. Και αν κάτι αλλάξει στην εμπορική πολιτική, στη γεωρική πολιτική, ή σε φρούτα, γάλα, τέφλα, κάτι, κάτι αλλάξει λοιπόν, στην πολιτική πολιτική, τότε έχουμε πολύ σοβαρές συνέπειες για αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει εκεί η σε φρουτα γαλα τεφλα κατι κατι αλλαξει στην μολική πολιτικη τοτε εχουμε πολυ σοβαρες συνεπειες για αυτους τους ανθρωπους ολα αυτα ειναι πολυ σημαντικα γιατι θα πρεπει να δουμε πως θα γινει εκει η αναπτυξη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ενδιαφέρουσες οι ευκαιρίες τέτοιας ενέργειας, ακόμα και από τα κύματα μπορεί να έχουμε ενέργεια από τα κύματα, τον ήλιο, τον άνεμο, σε πολλές από αυτές τις περιοχές μπορούν να έχουν αυτάρκη αυτά τα μέρη. Να είναι λιγότερο εξερτημένα από πλευράς ενεργείας. Με μεγάλη προσοχή όλα. Relancé par cette autre question. Par le passé, vous avez critiqué στο παρελθόν έχετε ασκήσει κριτική στην ε, Τρόικα, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και τις πολιτικές τη. Θα ήσασταν έτοιμοι τώρα λοιπόν να αλλάξετε λογική, να ε, μην ακολουθήσετε δηλαδή τη λογική της λιτότητα. γιατί ξέρετε ότι έτσι διαβρύνονται οι ανισότητες. Απάντηση. Πράγματι, άσκησα κριτική στην υπερβολική προσαρμογή που ζητήθηκε από τις χώρες αυτές, από την Τρόικα. Και συζητήθηκε και στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό το θέμα. Νομίζω πλέον να αναγνωρίζετε ότι ήταν υπερβολική αυτή η προσαρμογή. αντιληφθήκαμε ότι ένα κοινό νόμισμα χρειάζεται άλλου είδους εργαλεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε μια ελπίδα για τις περιφέρειες αυτές να βρουν δηλαδή ε, το δρόμο προς τη σύγκληση με τρόπο λιγότερο δυνηρό από ό,τι κατά το παρελθόν. Θα πρέπει να δούμε και την προσαρμογή του μηχανισμού αντιστάθμισης. Χρειαζόμαστε βράχοι πρόθεσμους μηχανισμούς σταθεροποίησης. Θα δούμε κατά πόσον κατατεθεί νέα πρόταση στο μέλλον. Και για το βραχυπρόθεσμο επίπεδο, γιατί και αυτό χρειάζεται στην Ένωση. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Αντζέλικα Μοτστανόφσκα. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι, αλλά δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη. Άρα δεν είναι δυνατό να αλλάξουν οι στόχοι και οι πολιτική. Αυτό που είπατε για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή, ότι πάνε χέρι-χέρι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε παρόλα αυτά ότι η χρηματοδότηση στις στοχές χώρες ε, έχει υποστεί πολύ μεγάλες ε, περικοπές. 23 για την Πολωνία, 7 για την Γερμανία για παράδειγμα, της 100. Ε, και επίσης υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών. Αν πιο στοχές χώρες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα κονδύλια, θα επιβραδυνθούν και οι πιο πλούσιες χώρες στην ανάπτυξή τους. Οι δημοσιονομικές αυτές προοπτικές ε, περικοπές θα οδηγήσουν τελικά σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή όχι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η οχι ευχαριστω παρα πολυ κοιταξτε θεωρω οτι η ερωτηση σας ε, έχει ένα στοιχείο το οποίο εξυπονοείται, δηλαδή το πώς διανέμονται τα διαρθρωτικά κονδύλια στις ε, διάφορες χώρες. Και κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι ε, τύποι, θα έλεγα, που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι είναι λογικοί. Δηλαδή, αν μια χώρα αρχίσει να αναπτύσσεται, χάνει την πρόσβαση σε κάποια κονδύλια. Και ε, όταν έχουμε μια χώρα που έχει προβλήματα να στηρίξει τις ε, περιφέρειές της. Υπάρχουν ε, προβλήματα γενικότερα με την ανάπτυξη και τις δουλειές. Οπότε ε, πρέπει η συνταγή, αν θέλετε, να βελτιώνεται συνεχώς και ο τύπος, και να διορθώνεται, αλλά προσπαθεί να επιτύχει μια αναλογία δεδομένη της ε, κατάστασης κάθε χώρας. Οπότε το Ταμείο δεν υπάρχει εκτός των ε, κανόνων. Οι αλλαγές οφείλονται στον ρυθμό ανάπτυξης της ε, κάθε χώρας. Παραδείγματο η Πολωνία τα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχει επιτύχει την σύγκληση και αξίζει συγχαρητήρια. Αλλά καθώς το επιτυγχάνει αυτό, ε, λογικό είναι ότι θα λαμβάνει λιγότερα. Το ίδιο συνέβη και στην Πολωνία, στην ε, Πορτογαλία, με συγχωρείτε, και αλλού. Οπότε τα κονδύλια πηγαίνουν ε, κατά προσήμιση και κατά κύριο λόγο στις χώρες εκείνες που ακόμα έχουν πολλή απόσταση να καλύψουν. Οπότε είναι θέμα το οποίο εξαρτάται και από την πορεία που ακολουθεί κάθε χώρα. Βεβαίως ε, ο κάθε τύπος ε, έχει τα όρια του. Δηλαδή όταν οδηγούμαστε σε μεγάλη μείωση τη χρηματοδότησης κάπου θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα συνολικά κοσά. Δεν μπορούμε ε, απλά να συγκρίνουμε την τωρινή περίοδο με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γιατί όταν μια πολιτική είναι επιτυχής, μετά οδηγεί πράγματι σε μείωση τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω άλλη μια ερώτηση πολύ σημαντική. Υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός σε επίπεδο Συμβουλίου και διαπραγματευθήκαμε τη δυνατότητα ε, διενέργειας κάποιων σχεδίων υποστήριξης φυσικού αερίου η αγορά συνδρομικού εξοπλισμού, χρηματοδότηση ε, αεροπορικών υποδομών. Συμφωνείτε ή με το Κοινοβούλιο ή όχι σε αυτή την προσέγγιση. Απάντησα ήδη σε μια ερώτηση για αεροδρόμια. Η τρέχουσα κατάσταση είναι εξή. Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων όπως τις εξόφως από μακρισμένες περιοχές, τα αεροδρόμια δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται. Γιατί είναι αντίθετα με το γενικότερο στόχο της σταδιακής μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη οικονομία στην Ευρώπη. Οπότε είναι ε, δυνατόν βεβαίω να φτιαχτούν αεροδρόμια, αλλά αυτό το οποίο δεν θα έχει κανείς θα είναι στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για τις επιπλέον εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε έτσι έχουν οι κανόνες αυτή τη στιγμή βεβαίως. Κατά περίπτωση ε, πρέπει να δούμε το πώς εφαρμόζεται στην ε, πράξη η αρχή. Σας ευχαριστώ. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση, λέει ο Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω πως δεν είναι υποχρεωτικό να επανέλθετε με δεύτερη ερώτηση και πρέπει να έχει σχέση με την αρχική ερώτηση επίσης. Τον λόγο έχει η κυρία Σιμών Σμιτμπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία υποψήφια επίτροπε, σε κάποια κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες τάσεις αποκέντρωσης στην λήψη αποφάσεων που πηγαίνουν από το κράτος στις ε, περιφέρειες. Ταυτόχρονα σε άλλα κράτη-μέλη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, η τάση συγκεντρωτισμού. Λοιπόν, για να γίνει αισθητή η περιφερειακή πολιτική σε όλες τις περιφέρειες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να βρεθούν εταίροι, τοπικοί, περιφερειακοί και κοινωνικοί οι οποίοι θα εμπλέκονται στην διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει στη ζωή αυτή η αρχή των εταίρων. Εδώ πέρα βεβαίως δυστυχώς ε, υπάρχει αντίσταση του Συμβουλίου όπου επιθυμεί κάπως πολύ πιο γενικόλογες διατυπώσεις. Οπότε το ερώτημά μου προς εσάς είναι το εξής. Εσείς ως Επίτροπος θα ενθαρρύνετε στο μέλλον τα κράτη-μέλη να δώσουν σταδιακά την διαχείριση των κονδυλίων συνοχής από το κεντρικό κράτος της ε, περιφέρειας ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σημαντική ερώτηση. Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να σεβαστώ τις ε, επιλογές που κάνουν οι χώρες εάν ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα ή ένα έργο το οποίο είναι περιφερειακό, τότε πράγματι πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο αρμοδιότητας και ευθύνης. Σκέφτομαι τη δική μου τη χώρα, πολύ συγκεντρωτική. Δεν είναι ερετές περιφέρειες, αυτή είναι μια επιλογή που ε, έχει γίνει στο εθνικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμβαίνει στην εσωτερική οργάνωση των κρατών. Έρχομαι λοιπόν στην επόμενη ερώτησή μου. Για να μπορέσει η πολιτική συνοχής ε, να λειτουργήσει και να λειτουργήσει αυτή η αρχή της εταιρική ε, σχέσης ε, χρειάζεται εμπιστοσύνη και εσείς είπατε στην αρχή σας δήλωση πως θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχουν ε, στην ε, συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ε, συγκρουόμενα συμφέροντα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή αναφέρομαι. Ο σύντροφός σας είναι αρμόδιος στην Πορτογαλία για την διανομή ακριβώς των κονδυλίων συνοχής. Υπάρχουν εδώ πέρα συγκροώμενα συμφέροντα ή όχι. Θα απαντήσω αγγλικά λέει η κυρία Φεραίρα, για να καταλάβουν όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να εξηγηθώ. Ε, αυτό σχετίζεται με την πρώτη μου απάντηση. Στην ε, Πορτογαλία δεν υπάρχουν περιφέρειες ως περιφέρειες, υπάρχουν διοικητικές μονάδες. Ο σύζυγός μου είναι καθηγητής ε, του Πανεπιστημίου, οικονομολόγος και ε, εδώ και τρία χρόνια υπηρετεί έναν από αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς ε, που ασχολείται ακριβώς ε, με την διανομή των κονδυλίων στην Βόρεια Πορτογαλία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων, καθώς αυτός είναι υπόλογος στον Υπουργό της κεντρικής κυβέρνησης, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τον ε, σχεδιασμό. Ότως και άλλως επειδή με ανησυχεί πάρα πολύ και το πώς φαίνεται η εικόνα αυτή. Είμαι πεπισμένη ότι δεν υπάρχει ε, κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Πρόκειται για δημόσια υπηρεσία, ε, ούτως ή άλλως δεν ε, είναι κάτι, μια ιδιωτική εταιρεία. Έγραψα όμως ε, μια επιστολή στην Πρόεδρο, την προταθήσα της Κομισιόν, ότι εάν κάποια στιγμή, ανα πάσα στιγμή, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, σας διαβάζω τώρα την επιστολή που έγραψα, θα λάβω οποιοδήποτε μέτρο για να μην υπάρχει και η εμφάνιση, η εικόνα οποιασδήποτε τέτοια σύγκρουση, Δηλαδή θα απέχω από οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων που αφορά τέτοια κονδύλια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα ή έμεσα τα προσωπικά συμφέροντα του συζύγου μου. Οπότε αν υπάρχει κάποια προσωπική πτυχή εγώ θα απέχω πλήρως Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορώ να λάβω απόφαση επί ενός τέτοιου θέματος και η ε, πρόεδρος της Κομισιόν θα αποφασίσει ή θα το αναθέσει σε κάποιον άλλον. Είμαι πεπισμένη ότι δεν θα συμβεί αυτό. Είμαστε ένα σύστημα που έχει κανόνες. Ο σύζυγός μου ποτέ δεν ε, συναντήθηκε ή δεν διαπραγματεύθηκε με τον προηγούμενο επίτροπο. Ούτε λήφθη κάποια απόφαση που τον επηρέαζε. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω Γι' αυτό απέστειλα αυτή την επιστολή προς την ε, πρόεδρο την επιλεγήσα της ε, Κομισιόν και όπως σας είπα είμαι έτοιμη για οποιαδήποτε μέτρα θεωρηθούν αναγκαία. Αυτή, αυτός είναι ο συμβιβασμός μου και το λέω δημόσια. Σας ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ την... Ευχαριστούμε και τη συνάδελφα και την Επίτροπο. Την υποψήφια Επίτροπο. Γιατί ήταν ειλικρινής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την ε, Επίτροπο για την πρόταση. Πώς θα εξασφαλίσετε να ε, είναι σε ετοιμότητα η Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή και δεν θα μείνει πίσω καμία περιφέρεια γιατί υπάρχουν κάποιες που θα πρέπει να έχουν κάποιες ευφύς ε, εξειδικεύσεις για να μπουν σε αυτήν την καινούργια φάση. Και πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα τα ταμεία θα βοηθήσουν τώρα που θα έρθει ε, η στρατηγική ή ε, σχετική, πώς θα θωρακίσετε την αναπτύξη όλων των περιφερειών, ακόμα και των μη προνομιούχων επίσης. Υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ δημοκρατίας, δημογραφίας και του δικού σας χαρτοφυλακίου. Τι γίνεται με την Ήπεθρο, τι γίνεται με τους αεροκατοικημένους τόπους πώς θα συνεργαστείτε με τους συναδέλφους με τα άλλα χαρτοφυλάκια, τι θα κάνετε και αυτά τα προβλήματα που θα είναι κρίσιμα όταν έρθει η ώρα της ψηφιοποίησης και καινοτομίας. Ε, Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που φίξατε. Αυτό που επιδιώκουμε την πρότασή μας είναι το εξής. να δούμε πώς θα πετύχουμε δύο πράγματα. Και τους δύο στόχους μας. Πιο ευφύ Ευρώπη, πιο καινοτόμα οικονομία, περισσότερη τεχνολογία και οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές να μην μείνουν πίσω και να καθυστερήσει η ανάπτυξή τους. Αυτό είναι ο ένας στόχος. Ο άλλος είναι ο εξής πιο πράσινη Ευρώπη, πιο συμβατή με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Έχουμε αυτό που λέμε θεματική συγκέντρωση. Δηλαδή, για κάθε κατηγορία περιφέρειας υπάρχει ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο για αυτά τα δύο θέματα που θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, ακόμα και στις πιο φτωχές χώρες, οι πιο φτωχές περιφέρειες, ε, κοιτάμε τι γίνεται σε κάθε επίπεδο, πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυσκολίες, πού υπάρχει δυσκολία χρηματοδότησης και έτσι προσπαθούμε να δούμε με τι επενδύσεις μπορούμε να πάμε ε, να πετύχουμε τους στόχους. Οπότε, είναι θέμα τυπολογίας, ας πούμε, χαρακτηρισμού της κάθε περιφέρειας και δεν θέλουμε να έχουμε κάποιους κατάτμιση. Αλλού να έχουμε καινοτομία και αλλού τίποτα. Προσοχή. Οι κεντροκατευθυνόμενες πολιτικές θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις επιπτώσεις επιτόπου. Οι στατικές επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να προσανατολίζονται στα πιο αναπτυγμένα μερικά της χώρας. Πολύ ενισχυτικό είναι όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και αυτό θα το λάβουμε υπόψη και θα λάβουμε όπως ακριβώς αυτό το, το, το, το παράγοντα της, ε, της επίπτωσης στη χώρα. Όμως μας, ε, ε μας ανισχύει, λέει κύριε Περιστό, τι γίνεται με τη χρήση των ε, πόρων. Δεν μπορούν να προωθήσουν και να εκτελέσουν τα βασικότερα πια. πιο βασικά προγράμματα για υποδομές. Εσείς τι θα κάνετε για αυτές τις περιοχές. Πώς θα αξιοποιηθούν ε, όπως ας πούμε για καινοτομία αυτή η πορεία και τι προτείνετε. Πώς θα είναι πιο αποτελεσματικά. Πώς θα πιάσουν τόπο τα χρήματα. Τεχνική αρρωγή ή τι. Για την χρήση των πόρων. Επίτροπος. Αυτό που ρωτάτε είναι θέμα ποιότητας θεσμών. Τι θεσμικές δομές υπάρχουν, ε, πώς είναι ο κοινωνικός ιστός, ας το πούμε, της ε, κάθε χώρας του κάθε τόπου, της κάθε περιφέρειας. Οπότε όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Πώς θα δώσουν τεχνική βοήθεια και έτσι τα προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά. Ναι, ανάπτυξη αλλά όχι με κάθε τίμημα. Περιβαλλοντική ανάπτυξη. Χρήσιμη, βιώσιμη. Νέες τεχνολογίες με την ανάπτυξη. Υπάρχουν περιθώρια στην πρότασή μας, ούτως ώστε όλα αυτά να καλυφθούν. Να βρεθεί η σωστή δοσολογία, η σωστή συνταγή και να έχουμε κερδισμένους τους πάντες εμπιστευτούμε τους τοπικούς παραγόντες και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι ότι προγράμματα τρέχουν ε, τους ε, βρίσκουν όλους κερδισμένους και έχουν βιωσιμότητα. Ο επόμενος. Καλώς ορίσατε, Επίτροπε. Εδώ, εδώ είμαι, λέει η κυρία Νταμάτου. Το Μάρτιο περάσαμε ένα κείμενο και είπαμε ότι θα πρέπει να έχει για την εθνική συγχρηματοδότηση, για το σύμφωνο σταθερότητα να βοηθήσει περισσότερο. Βλέπετε με περισσότερη ευελιξία λοιπόν και σήμερα μα είπατε ότι στη Νέα Επιτροπή θα γίνει σχετική συζήτηση και θα αναθεωρήσετε κάποια κριτήρια για το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Πάρα πολύ λεπτό, ευαίσθητο το θέμα. Τι θα γίνει με την ε, απασχόληση, την ανάπτυξη τη λιγότερο προμήθειε περιοχές. Το επιβεβαιώνετε αυτό που υποσχεθήκατε. λόγω του ελλείμματος θα βγουν οι εθνικές χρηματοδοτήσεις για το περιβάλλον, για την αλληλεγγύη του κλίματος. Θα προχωρήσετε παραπέρα όσον αφορά τις ε, ενισχύσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να κάνετε για, αυτό, για την εθέρωση αυτού του πλαισίου διάλογο με το Συμβούλιο. Eh, muito obrigada. Eu eh, o que disse é que assuntos como esse têm de ser tratados. Eh, ευχαριστώ. Όπως είπα, ε, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Γίνεται εδώ πέρα μια ανάλυση του θέματος, αλλά δεν είναι υπό την ηγεσία μου. Πολλά από αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά είναι μια διαδικασία περίπλοκη και μακροσκελής και απαιτεί και συναπόφαση. Και είναι και θέμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτά λοιπόν είναι αρμοδιότητες ε, του συναδέλφου που είναι αρμόδιος για την οικονομία. Και άρα ε, εγώ σας εγγυώμαι ότι θα είμαι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση και θα προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση στο πακέτο, αλλά δεν μπορεί να αγγίθω τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δυστυχώς ε, όλα αυτά συνδέονται με το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξη. Πώς θα έρθετε πραγματικά σε επαφή με περιφέρειες και δήμους που έχουν περιορισμένη διοικητική ικανότητα. Υπάρχει κάποια τεχνική αρρωγή που δίνεται, αλλά δεν επαρκεί. Οι δήμοι δεν μπορούν να ε, τρέξουν τέτοια έργα, αλλά από την άλλη δεν μπορούν και να τα συγχρηματοδοτήσουν λόγω του Συμφώνου Σταθερότητας. Σας ε, ευχαριστώ. Ε, έχει πολλά μέρη η ερώτησή σας. Έλεγχοι. Χρειάζονται έλεγχοι. Υπάρχει μια ευθύνη για το ευρωπαϊκό χρήμα και είμαστε υπόλογοι στους πολίτες μας έτσι. Οπότε οι έλεγχοι χρειάζονται. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν στις προτάσεις της είναι να κάνει τα πράγματα πιο απλά, πιο ευανάγνωστα, ειδικά για τις μικρές εταιρείε και τους μικρούς δικαιούχους. Αλλά τούτου λεχθέντος πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Είναι μια τεράστια ευθύνη να διαχειριζόμαστε λεφτά που ανήκουν στους πολίτες μας. Τα πληρώνουν φόρους αυτά τα πράγματα, οπότε πρέπει να ενισχυθεί η ποιότητα. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε νέους μηχανισμούς που δεν προσθέτουν προσθέμενη αξία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει έλεγχος. Ξοδεύτηκαν σωστά τα λεφτά. Αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει και στην βελτίωση της ε, ουσίας. Ε, τα έργα πρέπει να ελέγχονται, αλλά πρέπει να υπάρχει αντίκτυπος ε, και στην περιφέρεια. Η δουλειά γίνεται, εντάξει, βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, οι προτάσεις συζητιούνται αυτή τη στιγμή, νομίζω θα βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα δώσω τώρα το λόγο στη Μαργαρίδα Μάρκες, που είναι μέλος Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Επίτροπε, υποψήφια. Ε, όλες οι χώρες της Ένωσης ε, λαμβάνουν χρήματα Τη συνοχή, αμέσω ή αμέσω. Η Πορτογαλία είναι μια χώρα όπου τα αποτελέσματα των κονδυλίων της συνοχής είναι πολύ ορατά. Όλοι ξέρουμε πως ε, έχετε έρθει εδώ πέρα σε μια ακρόαση για να γίνετε Ευρωπαίοι Επίτροπος, όχι υπουργό ε, τη Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία θα σεβαστεί το άρθρο 245 της ε, συνθήκη. Λοιπόν, στη νέα γενιά πολιτική συνοχή, ο στόχο τη συνοχή που είναι ιδρυτικό στόχο τη Ένωση, <laughs> πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Οπότε η χρηματοδότηση της συνοχής ε, πηγαίνει πολύ πέρα από το... τον φάκελο της χρηματοδότησης της συνοχής ε, της ίδιας. Οπότε θα ήθελα να γνωρίζω εάν η φιλοδοξία σας για το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής ε, είναι αναλογή και πρέπει να πω ότι χάρηκα που άκουσα ότι είστε ανοιχτοί στην συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν και για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει στο των δυνατόν για να έχουμε μια έγκαιρη συμφωνία για το ΠΙΔΛΤΑΠΗ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Πράγματι είναι ένα σχόλιο σωστό, επίκαιρο. Και βεβαίω ανταποκρίνεται και στις ε, ανησυχίε μας. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε έχει μια κάποια αστάθεια όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ίσως λοιπόν υπάρχει ανάγκη να πάμε να τα ξαναδούμε αυτά με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ίσως χρειαστεί να γίνουν αλλαγές και οπωσδήποτε και εγώ θα εμπλακώ ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω καλό θα ήταν να κινηθούμε πιο κοντά στις θέσεις του Κοινοβουλίου ευπρόσδεκτο οπωσδήποτε αλλά ε, δομικά θα έλεγα, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα των ίδιων πόρων. Υπάρχουν περισσότερες ανάγκες ε, όλο και πιο ποικιλόμορφες. Υπάρχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου που θα πιέσει πολύ τους πόρους. Η Κομισιόν είναι ένας τεχνικός φορέας και αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι πώς θα συνεισφέρουμε για να δημιουργήσουμε μια κοινή, κοινό αίσθημα ευθύνη ε, εντός της ε, Κομισιόν με τις δικές μας ε, εμπειρίες και διαφορετικές απόψεις βεβαίως. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όπως είδατε και στις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι το μέσο της ε, σύγκλησης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι συμπληρωματικό με τα άλλα μέσα και να προσθέτει κάποια προσθέμενη αξία, να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό κύκλο. Πώς μπορεί να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιβραδύνσεις στην οικονομία και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα και την σύγκληση, πώς θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα κριτήρια ε, διανομής για να επιδευτούν οι στόχοι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Μιλάτε λοιπόν προφανώς ε, για το μέσο αυτό το οποίο έχει ως στόχο την χρηματοδότηση των ε, διαρθρωτικών πολιτικών στα κράτη-μέλη. Μου αρέσει εμένα η λέξη διαρθρωτικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις γιατί μπορεί να παίξουν ένα θετικό ρόλο στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είτε του στήματος εκπαίδευσης ή της υγείας και όπως είπα στην αρχική μου τοποθέτηση ε, μπορεί να είναι το πώς διαχειρίζεται κανείς ε, τα δάση για να προλάβουμε ε, καταστροφές, π.χ. δασικές πυρκαγιές. Οπότε το σκεπτικό είναι ότι θα μπορούμε να στηρίζουμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μην περιορίζουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από το ότι δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο. Αλλιώς ε, δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις ε, πολιτικές τηρώντας ταυτόχρονα το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής. Βεβαίως ε, το μέσο αυτό βασίζεται στις εμπειρίες της προηγούμενης θητείας της Κομισιόν όπου υπήρχε μόνο τεχνική αρρωγή, δηλαδή χώρες που έκαναν προσπάθεια για να ενταχθούν στο κοινό νόμισμα βλέπουν τώρα ότι υπάρχει και ένα παρόμοιο σύστημα για τις μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίδια Περέρα από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η περίοδος οικονομικής ανάπτυξης είναι ευκαιρία για διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η εκλογική περίοδος ουσιαστικά ε, βάζει σε πειρασμό τις κυβερνήσεις να αναστρέψουν αυτή την τάση. Είδαμε τις πολιτικές λιτότητας που σε Ελλάδα, Πορτογαλία και άλλες χώρες ε, δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Και οι μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης επίσης δεν έχουν προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, ο Ρονάλντο δεν έχει βάλει ένα γκολ. Άρα ούτε στην Ευρωζώνη ούτε πουθενά αλλού έκανε ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Πώ λοιπόν θα μεταρρυθμιστεί η οικονομία, πώ θα μεταρρυθμιστεί το ευρώ. στι γραπτέ σα απαντήσει μιλάτε για τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και λέτε ότι είναι προπόθεση για όλα. Για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, μα δεν δίνεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε όμω πρέπει να ξέρουν συγκεκριμένα για ποιε μεταρρυθμίσεις μιλάτε, τι θέλετε να αλλάξει, για παράδειγμα στην αγορά εργασία ή στα σχολεία, στα νοσοκομεία απάντηση. Με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω. Αλλά αφήνω κατά μέρος ε, τα σχόλια για την εσωτερική πολιτική. Έρχομαι στους στόχους μου. Ποιοι είναι οι στόχοι μου. Δεν είναι δικοί μου στόχοι βέβαια. Ε, ε, στην ουσία κάθε χώρα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να κάνει διαπραγμάτευση και να τα συζητήσει όλα αυτά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. προσπαθώντας να δει από αυτές τις πολιτικές που εντοπίστηκαν, ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ουσιαστικά για αναδιοργάνωση πρόκειται, αλλά και για επενδύσεις στο κοινωνικό επίπεδο κυρίως. Και θα πρέπει κάθε χώρα να ορίσει τη δική της στρατηγική. Δεν επιβάλλονται, και αυτό είναι σημαντικό τέτοιο τις πολιτικές, είναι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο των συστάσεων αναχώρα, αλλά οι χώρε θα πρέπει να προτείνουν το χρονοδιάγραμμα και πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Ε, επερώτηση. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Το σχόλιο μου δεν αφορά στην πολιτική. Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά τις διαρκτικές μεταρρυθμίσεις. Είπατε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά ανά χώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι την ίδια γραμμή θα ακολουθήσει η Κομισιόν. Πρέπει να έχει κάποιο γνώμονα, κάποια γενική κατεύθυνση. Έτσι είναι τα πράγματα. Ελπίζω αυτό να απαντήσετε και σε ό,τι αφορά τη σύγκληση. Υπάρχει ο περιπολισμός στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ένα φιλοευρωπαϊκό όραμα, αλλά φαίνεται να εξανεμίζεται λίγο και να δημιουργούνται μίνι τρόικες. Μία για την αγορά εργασίας, μία για την παιδεία, μία για την υγεία. Έτσι είναι τα πράγματα και αυτή είναι η φιλοδοξία σας. Για τον προβληματισμό της Ευρωζώνης. Αλλιώς δώστε μας κάποιες ε, λεπτομέρειες παραπάνω γιατί άλλως θα φύγουμε με πολύ μεγάλη απογοήτευση από εδώ μέσα απάντηση. Ακούστε, αυτές οι μικρές τρόικες, ε, τροικούλες, δεν ξέρω πώς να τις πω, θα μπορούσαν να είναι και πρόοδος, ξέρετε. Τέλος πάντων. Αφήνοντας κατά μέρος τα εγώ αγωνίστηκα πολύ κατά της Τρόικας, αλλά τα πράγματα αλλάζουν, έχουν αλλάξει πολύ στην Ευρώπη. Έχει αλλάξει και ο οργάνωση των οικονομικών πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, κατά την άποψή μου, θα βοηθήσει να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, ε, ποιε ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της χρήσης του ενίου νομίσματος. Βέβαια, οι χώρες είναι αυτέ που επαναλαμβάνω θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Και εκεί μπαίνει μετά η Τρόικα. Ποιο είναι το πρόβλημα με την Τρόικα. Ότι επειδή η Ευρώπη δεν είχε παρκώ ξεκάθαρε δομές, δημιουργήθηκε αυτή η δομή που κατά την άποψή μου δεν λειτουργήσε. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε το six pack, έχουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και μία δέσμη προτάσεων. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένες προτάσεις, σας παραπέμπω στις ειδικές τάσεις αναχώρα. και στις μεταρρυθμίσεις, τις εθνικές, το σχέδιο δηλαδή μεταρρυθμίσεων της κάθε χώρας. Υπάρχει και το παράρτημα D, δέλτα, που υπάρχει ένα συγκεκριμένο κατάλογο ε, με τα είδη των έργων και σχεδόν που θα πρέπει να φέρουν σε πέρα οι χώρε. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει οι χώρε να κάνουν τι επιλογέ του και να πούν τι θα κάνουν συγκεκριμένα. Να μην ασκούμε μόνο κριτικέ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα προ τα εμπρό. Ζωζέ Κουσμάου έχει τώρα το λόγο, μέλος Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και Επίτροπε. Μας εξηγούσατε ότι έχει αλλάξει πολύ η οικονομική πολιτική, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ναι, γίνεται κουβέντα για επενδύσεις, αλλά τι πάει να πει επενδύσεις υποβοήθηση στην ανάπτυξη, αλλά τι γίνεται με την αναδιανομή, τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την χρηματοδότηση συνοχής. Λέμε ότι θα υπάρξει κάποια υποστήριξη, αλλά εσείς χέρι με χέρι με το Κοινοβούλιο θα αγωνιστείτε για να μην υπάρξει καμία περικοπή στην πολιτική συνοχής. Στο χειρότερο σενάριο. Και θα συμφωνούσατε ότι χρειάζονται επενδύσεις κατά της φτώχειας και της ανισότητας ε, για το κλίμα, για τις ε, κρατικές υπηρεσίες και όλα αυτά να μην κολοβώνονται από τους κανόνες για το έλλειμμα. Να σας απαντήσω με μεγάλη μου ευχαρίστηση, λέει η κυρία Φερέρα. το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Σύμφωνο Σταθερότητας έχουν κάνει βήματα πρόοδο. Δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια και ρόδινα. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βήμα-βήμα χτίζεται η Ευρώπη. Θα πρέπει να βελτιωνόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας και λοιπά. Ε, τα άλλα που ρωτήσατε, νομίζω ήδη τα έχω απαντήσει. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει συνεχώς να κολλάμε σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν ε, σενάρια περικοπής ε, από τον προϋπολογισμό. Εάν οι αρχές του προϋπολογισμού βάλουν ένα πιο ψηλό ταβάνι, αν όριο, εντάξει. Θα πρέπει, συμφωνώ, να προστατεύσουμε την πολιτική συνοχής. Και ιδίω να προστατεύσουμε την γεωργία. Χρειάζεται μεταρρύθμιση και στη Γεωργία, χρειάζεται χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχή. Αυτά όλα είναι σημαντικά για την Ήπεθρο. Θα πρέπει να έχουμε αρκετές, αρκετούς πόρους, να αντιμετωπίζουμε τα εκάστοτε προβλήματα, οπότε και εγώ θα αγωνιστώ για αυτά τα θέματα που είναι του δικού μου χαρτοφυλακίου. Αλλά θα πρέπει να αναζωογονηθεί και η εσωτερική αγορά, ιδίω μια που έχουμε κοινό νόμισμα. Βέβαια κάθε οικονομία έχει άλλους ρυθμούς και αυτό κάνει τα πράγματα δύσκολα. Ξέρουμε τι γίνεται στην πράξη. Έχουμε δηλαδή πολλή δουλειά μπροστά μας. Ο επόμενο. Όχι, επέρατε. Και τι έγινε, για να δω, πώς λειτουργήσε το πράγμα. Κάποιοι κανόνες τηρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ε, περιθώριο ελιγμών, οι άλλες χώρες δεν έχουν, οπότε είναι στριμωγμένες οι Άρα, τι εννοούμε όταν μιλούμε για μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας, τι είναι, μία από τα ίδια απορρίθμιση στην αγορά, περικοπή ε, δημοσίων κοινοφιλών υπηρεσιών, τι γίνεται, περικοπή στην περικοπή, επίσης αν ξέρετε τι θα πει υπεύθυνη η οικονομική πολιτική, εάν η Επιτροπή αναλάβει τις ευθύνες της και οι χώρες μας σε αποτέλεσμα των πολιτικών σας ξαναπέσουμε στην κρίση, τότε τι γίνεται. Δεν θα πρέπει να επιβάλλετε τις μεταρρυθμίσεις. Άρα εσείς υπόσχεστε ότι θα αρνηθείτε περικοπή στα διευθυντικά ταμεία. Δηλαδή να μην έχετε χρηματική κύρωση, οικονομική κύρωση, εάν κάποιος δεν πληρεί τα όσα διατάσσει κομισιόν. Κοιτάξτε, τι θα πει συνοχή. Ε, είναι κάτι που διέπεται από κάποια νομοθετήματα, είναι θέμα επίσης ε, ερεσιμότητας μακροοικονομικής και όπως λέμε σήμερα έχουμε κάποια μέτρα για να μετριάζουμε αυτά τα φαινόμενα Άρα, με γνώμονα αυτά θα προχωρήσουμε. Εγώ λαμβάνω υπόψη ε, τα όσα θέλει το Κοινοβούλιο Και κατά τη γνώμη μου, για τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να χαράξουμε κάποιες πολιτικές που οδηγούν σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των χωρών που το χρειάζονται. Όχι, δεν μπορώ όμως εγώ να το αποφασίσω μόνοι μου και τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να το κουβεντιάσουν. Ε, βέβαια και με υπέρ της Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε από την Οικονομική Επιτροπή. Λαμβάνουμε ότι δεν μπορείτε να μας πείτε ε, το τι θα είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αλλά ε, μπορείτε να μας πείτε ε, πότε θα συζητηθεί, πότε θα εφαρμοστεί. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, πώς θα διασφαλίσετε ότι το Ταμείο αυτό δεν θα περιοριστεί μόνο σε περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά θα καλύπτει και κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο, ειδικά στους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Δεύτερον, θα δεσμευτείτε ε, ότι δεν θα καταλήξει το νέο ταμείο σαν το εύση το οποίο θα καταλήγει σε μοχλευμένα ταμεία τα οποία θα πηγαίνουν στις περιοχές που αποδίδουν καλύτερα. Και τρίτον, όπως ε, ξέρετε, τα συμπεράσματα του Ιουνίου 2019 αναφέρουν ξεκάθαρα την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις, η κατάσταση του κάθε κράτους ε, μέλους. Θα παλέψετε το Ταμείο αυτό να στηρίξει τα νησιά και τις περιφερειακές περιοχές για να ξεπεράσουν ειδικά τις συνθήκες αυτές, ειδικά όταν μιλάμε για ε, μεταφορές και για καθαρότερα συστήματα ενέργειας. Κύριε Βουλευτά, σημειώνω την ερώτησή σας και την φιλοδοξία σας. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι ε, εντάξει δεν μπορώ τώρα να εικάσω εγώ ποιοι θα είναι οι συμβιβασμοί. Αλλά εργαζόμαστε πάνω στο θέμα. Κάνατε μία ερώτηση για το αν θα πρέπει το ταμείο αυτό να ασχοληθεί με τα ζητήματα των ε, νησιών. Εξαρτάται. Ε, κοιτάξτε, πρόκειται και για ένα ταμείο περιορισμένο. Μιλήσετε εδώ πέρα για 4,8 δισεκατομμύρια. Το ταμείο αυτό λοιπόν πρέπει να συμπεριληφθεί, να είναι πακέτο με τα ταμεία συνοχής. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν να διαρθρωθεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρότερα προβλήματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, αλλά πρέπει να δούμε τα ενοποιημένα μέσα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές καταστάσεις. Για την ώρα γνωρίζουμε, τα ήθελα να το διευρύνουμε κάπως, και θα δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να το μοχλεύσουμε αναφέρατε με αρνητικό τρόπο το, το σχέδιο Juncker, το παλιό πρόγραμμα Juncker. Πρέπει να δω αυτά τα μέσα γιατί δεν μπορούμε να καταγραμματίσουμε τα πάντα σύμφωνα με τα κονδύλια. Πρέπει να υπάρχει μια μόχλευση. Για τις κοινωνικές πτυχές εκεί μπορώ να σας απαντήσω οπωσδήποτε ναι πρέπει να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός, κάποια κοινή παρέμβαση η οποία με βάση τις περιφέρειες θα έχει το κοινωνικό ταμείο, την κοινωνική ένταξη, θα τα συνδυάζει όλα αυτά για να υπάρξει ανάπτυξη κάθε περιοχή. Αυτά και με συγχωρείτε. Ναι. Κάτι σχετικό λοιπόν όταν μιλάμε για περιφερειακές περιοχές και νησιά. Θεωρείτε ότι μπορούν να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των όσων θα θέλατε να κάνετε και της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης. Πολύ δύσκολη ερώτηση, δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα λεπτό. υπάρχουν κάποιες αιρέσεις, όπως ξέρετε, και εξαιρέσεις ε, όταν μιλάμε για τα νησιά στην πολιτική του ανταγωνισμού και για κάποιους λόγους ίσως πάλι να υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ε, στο θέμα αυτό. Ε, εξαρτάται από την κατάσταση την συγκεκριμένη, αλλά υπάρχει βεβαίως το προηγούμενο αυτό, ότι υπάρχουν εξαιρέσεις από την πολιτική ανταγωνισμού όταν ε, είναι ένα πολύ μικρό νησί που δεν μπορούμε να βρούμε ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός ε, εγγυημένα. Οπότε θα δούμε, θα συνεργαστούμε μαζί σας με το Κοινοβούλιο για να φτιάξουμε αυτό το μέσο, αλλά ας μην φτιάχνουμε έτσι απομονωμένες πολιτικές που θα κάνουν πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Um, Commissioner Designate. Κυρία Τζιλέβανς, ε, η, απο... η αποβιομηχάνηση είναι ένα πρόβλημα για πολλές περιφέρειες. Στην Ουαλία, την περιφέρειά μου, έχουμε μακρά εμπειρία οι δημοκρατικές αλλαγές επίσης επηρεάζουν στις αγωγικές παρατηρήσεις. Μιλήσατε για τους ε, νέους ανθρώπους, ε, τα νέα μυαλά τα οποία εγκαταλείπουν ε, για λόγους εκπαίδευσης ή απασχόλησης της πατρίδες τους και πόσο να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες και τους νέους, με ποιο τρόπο. Όλα αυτά υπονομεύουν την πρόοδο, υπονομεύουν τη συνοχή και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω θα έχετε στην ε, Κομισιόν μια ομάδα εργασία ε, ειδικών για να δει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ε, μειωθεί η φυγή των νέων από αυτέ τις περιοχές. Βέβαια, η δική μου περιφέρεια μπορεί να είναι εκτό τη Ένωση. και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω πώς θα εξασφαλίσετε τη συνεχή μας συμμετοχή στα δύο συνοριακά προγράμματα που είναι πολύτιμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φεραίρα. Είναι πολύ ε, κρίσιμο το θέμα που αναφέρεται. Ανεξαρτήτως της χώρας της περιφέρειας από την οποία προερχόμαστε, όλοι το ζούμε και θέλουμε να δώσουμε περισσότερη εκπαίδευση, κατάρτιση, να επενδύσουμε στους ανθρώπους. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες ως προς αυτό και βέβαια ε, δεν έχουν μετά καλούς μισθούς, οι και φεύγουν. Η φυγή κεφάλων Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερος. Ενστικτοδός θα έλεγα, ναι βεβαίως να δημιουργήσω μια ομάδα ε, εργασίας εμπειρογνωμόνων. Δεν ξέρω τώρα μήπως υπάρχει κάτι στις υπηρεσίες, στις αρμόδιες, ε, μπορεί να υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε κάποια γενική διεύθυνση. Πάντως θα το δω, θα το συζητήσω με το προσωπικό και θα δω τι γίνεται. Γιατί είναι μια ανησυχία που και εγώ συμμερίζομαι διότι αν χάσεις αυτούς τους ανθρώπους, βέβαια φυσικά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρουν μια απασχόληση που θα είναι ανάλογη με τα προσόντα τους. Πρέπει να υπάρχει δημόσια και πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων και επιχειρήσεων για τις περιοχές τις συγκεκριμένε που μιλάμε. Και πρέπει να είναι ένα πακέτο αυτό. Αλλιώς δεν λειτουργεί. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το μόνο που μπορώ να σας προσχεθώ αυτή τη στιγμή είναι ότι θα το μελετήσω πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ, κύριε Εύαν. Σε, σε συνέχεια θα μιλήσω για την ισότητα των φίλων και τη διάσταση του φίλου και τη συμπερίληψη της πολιτικές. Οι δεσμεύσεις σας ε, μας είναι πολύ καλό νέο σε μένα και στην ομάδα μου, αλλά στρατηγική σαφή για τη ισότητα των φύλων με συγκεκριμένους στόχους δεν υπάρχει ακόμη στο νέο πι Ούτε από ομαδοποιημένα δεδομένα υπάρχουν για το φύλ. Γιατί αυτό θα βοηθούσε να χαραχθούν και οι κατάλληλε πολιτικέ βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Επομένω, σα ερωτώ, τι βήματα θα κάνετε για να ε, συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου στην κατάρτιση του προπολογισμού για το επόμενο ΠΔΠ, το λεγόμενο gender budgeting. Κυρία Φερέρα, ναι βεβαίω, πολύ σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ που το θέσατε και επαναλαμβάνω ότι πράγματι με ενδιαφέρει και θα κάνω πάντο δυνατόν για να μπορέσουμε να ελοπίσουμε προγράμματα που θα έχουν αυτό το στοιχείο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θετικό πρόσφορο έδαφος και η ισότητα, η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων πιστεύω ότι μπορεί να ενταχθεί στις γενικές αρχές που ε, δημιουργούν πρόσφορο έδαφο σήμερα για τη διαχείριση των κονδύλων και των ταμείων. Και στη δική μου τη γενική διεύθυνση, εγώ ε, έχω δει το ανθρώπινο δυναμικό, μιλάω για τη ρέγγιο δηλαδή τώρα. Και στον πίνακα επιδόσεων, το scoreboard, γίνεται λόγος για τον υψηλό φόρτο εργασίας και την ανάγκη ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Και είναι μικρότερος ο αριθμός ε, των ε, γυναικών ε, στα ανώτερα στελέχη στη ΓΔΡ. Θα πρέπει να το δούμε λοιπόν εσωτερικά γιατί και καλυμμένα κατά κάποιο τρόπο, οι γυναίκες ε, αποχωρούν είτε ο θέλος όχι από την ανώτερη ε, διοίκηση. Και αυτό δεν είναι καλό. Στεφάν Μπιζού. Καλησπέρα σα, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Η Ευρώπη είναι γεμάτη από προκλήσει. Είναι ένα έδαφο με προκλήσει, αλλά και με πολλέ ελπίδε. Και αξιοπρέπεια απέναντι στην ε, ανεργία, ε, ασφάλεια απέναντι στην κλιματική απορρίθμιση, ελπίδα για την ισότητα των ευκαιριών πολύ απλά. Και δική μας πολιτική ευθύνη, συλλογική μας πολιτική ευθύνη είναι να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις αυτά στις θεμητές διεκδικήσεις και απαιτήσει των πολιτών από όλη την Ευρώπη. Ακόμη και αν απέχουν 10.000 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες, αν ζουν σε μια από απόκεντρη περιφέρεια, ε, στα γαλλικά ε, υπερπόντια εδάφη. Εκεί και αν πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά τη συνοχή και ζητώ ε, να υπάρξει αυτή η αποτελεσματικότητα που θα μεταφραστεί ε, με ένα τέτοιο αντανακλαστικό για τις ε, πολιτικές, περιβάλλον, υγεία, γεωργία, αλία πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις απομακρυσμένες περιφέρειες. Είπατε δεν θα αφήσετε κανέναν να μείνει πίσω, ε, δεν θα καταλήψετε κανέναν. Μας περιγράψετε ποια είναι τα κατεπήγοντα προβλήματα. Μπορείτε να δεσμευτείτε για μια μόνιμη επαγρύπνηση και για συγκεκριμένες δράσεις για τους πιο ευάλωτους και απομακρυσμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Κύριε Φερέρα, εύκολη είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ναι, φυσικά και δεσμεύομαι. Πραγματικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα είναι συλλογική ευθύνη, σίγουρα, και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Δεν είναι η μόνη βέβαια περίπτωση κεντρε. περιφέρειες. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που πρέπει να φροντίσουμε. Όμως, γενικώ πώ είναι κάπως πιο ιδιαίτερες από αυτήν την έννοια οι εξωξαπόκεντρες περιφέρειες. Σας ευχαριστώ για τη μέθοδο. Δυο λόγια αν μπορείτε να μας πείτε, η οργάνωση της δικής σας γενικής διεύθυνσης ε, και η σχέση σας με τους άλλους επιτρόπους και σε σχέση με τις που αναλάβατε. Μήπως θα μπορούσατε να έχετε μια τριμηνία πλατφόρμα μαζί με τους άλλους επιτρόπους, ίσως και με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να είμαστε εγκάρσιοι και αποτελεσματικότεροι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, θα την σκεφτώ θα δω. Θα συζητήσω με τις υπηρεσίες. Και ίσως βρούμε μια λύση. Αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει αυτό που λέτε, όπως ακριβώς το λέτε. Πάντως θα το αναλύσω πολύ σοβαρά. Merci. La parole à notre cher collègue José Manuel Fernandez, membre de la Commission. José Manuel Fernandez, ο αγαπητός συνάδελφος από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψηφία Επίτροπε, ικανότητες, φιλοδοξία, θάρρος, αυτά είναι. Και υπ' αυτού του όρου, άλλοι τα πήγαν καλά από του επιτρόπου και άλλοι όχι. Ο κ. Μέντε απέσπασε 80 εκατομμύρια για την έρευνα. Με πρόταση 100 εκατομμύρια μετά 20 5% αύξηση, αλλά η Επιτροπή ανταυτού πήγε σε περικοπές. 1,6 δις περικοπές δηλαδή στην Πορτογαλία. Αυτά πώς να τα χωνέψουμε. Πάντως το ίδιο το Ταμείο Συνοχής αποσκοπεί στο να καλύψει τις φτωχότερες χώρες. Στην πρόταση της Επιτροπής όμως προβλέπεται περικοπή 45% που είναι απαράδεκτο. Εσείς τι λέτε. Είναι δυνατόν έτσι να τη λέμε αυτή την πολιτική, πολιτική συνοχή. Αυτό το μείον 45% δεν αφήνει περιθώριο για καμιά συνοχή. Άρα ποιο είναι το καλύτερο σενάριο. να συνεχίζει η συνοχή να είναι προτεραιότητα. Στις έγγραφε απαντήσεις είπατε ότι το καλύτερο δυνατό σενάριο υπάρχει, δηλαδή το να γίνουν περιορισμένες περικοπές. Άρα τι, παραιτηθήκαμε τι προσπάθειες. Έτσι θα αποδυναμωθεί και η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ, λέει Ένα σωρό συνάδελφοι το ερώτησαν και ήδη απήντησα Απήντησα σε όλους. Συνεχίζετε να μου λέτε τα ίδια. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί καλή αφετηρία. Και αν η μόνη εναλλακτική είναι να απορρίψουμε την πρόταση, τότε θα επεξεργαστούμε ξανά αυτήν. Άρα θα το ξαναδούμε για τις διαπραγματεύσεις. Ε, βέβαια και θα γίνουν τριμερείς διάλογοι και είμαι βέβαιος ότι αύριο θα έχουμε επίσης επαφές στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται να εξελίξει. Να δούμε πώς να εξαντλήσουμε τα όρια του προϋπολογισμού. Μίλησατε για την Πορτογαλία. με το πόσο κακές αυτές οι περικοπές, αλλά σας υπενθυμίζω, μήπως και το ξεχάσαμε, ότι έχουμε σήμερα μείωση 7% των σχετικών τιμών. Και όταν περάσαμε από το σύστημα του 13-16 μέχρι 14-20 είχαμε μείωση και περικοπή 10,5%. Και είπατε ότι έχουμε 1,6% λιγότερο για την Πορτογαλία. Όμως την τελευταία φορά είχαμε περικοπή 2,3% στην Πορτογαλία. Άρα δείτε το σύνολο της εικόνας. Ε, τώρα έχουμε τον Brexit. Τελευταία φορά που τα είπαμε, τα πράγματα δεν ήταν τόσο φορτισμένα. Τώρα όμως έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε αυτή τη συγκυρία και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Φυσικά και πάρα πολύ καλά τα είχε πάει ο Μουέντε, δεν θα κάνει όμως σήμερα. Το 2014 που συζητήθηκαν οι δημοσιονομικές προοπτικέ, τα πράγματα ήταν πολύ πιο ρόδινα. Είναι δεδομένο το τι θέλουμε. Ε, δεν βγαίνει τίποτα με το να επιμένουμε στα ίδια. Ελπίζω με το Συμβούλιο θα τα διαπραγματευτούμε καλά. Πάντα πάντα να υπολογίζετε στη βοήθεια από εμά και από μένα προσωπικά. Φέρναντε ξανά. Ναι, ναι. Με διορθώσατε. «10% ήταν και πάμε τώρα για άλλο ένα 7% ως περικοπές. Ε, αφού δεν συμφωνήσατε με την πρώτη περικοπή, γιατί θέλετε τη δεύτερη, γιατί συμφωνείτε με τη δεύτερη. Τι γίνεται με τον τύπο κατανομής. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί. Μερικές χώρες που είναι πλούσιες παίρνουν περισσότερα και κάποιες άλλες που είναι φτωχότερες παίρνουν λιγότερα με τις ε, περικοπές. Επίτροπος, σας το ξεκαθαρίζω, δεν συμφωνώ με καμία περικοπή. Ούτε παλαιότερα συνεφώνησα, ούτε τώρα. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω πώς είχε τότε η κατάσταση. Ε, βέβαια δεν συμφωνώ. Καμία περικοπή. Είπατε κάτι για τον τύπο κατανομής, τον τύπο Βερολίνου. Είναι περίπλοκος, Δεν τον έβγαλα εγώ. Το 2000 συζητήθηκε το θέμα της ε, ευημερία σε εθνικό επίπεδο. Ε, είναι λίγο απλουστευτικό να τα λέτε έτσι. Δεν μπορούμε τώρα να κατεβάσουμε το κεφάλι μας άλλο τύπο. Κάποιες χώρες ε, έχουν λιγότερη περικοπή, όμως αναπτύχθηκαν, προόδευσαν, υπάρχει πρόοδος και αυτό και θέλουμε. Οπότε καταρχήν αυτές οι χώρες ε, επειδή προόδευσαν δεν παίρνουν αρκετά ε, από αυτά τα κονδύλια. Αλλά αυτό που το οποίο χρειάζεται φυσικά είναι η σύγκληση ο Πρόεδρος. Ωραία έγκληση και αυτός ο γύρος των ερωτήσεων και... Κύρια υποψήφια επίτροπε, μπορείτε να προβείτε σε μια σύντομη δήλωση και έτσι να ολοκληρώσουμε. Έχετε πέντε λεπτά και θα λάβει ο υποφαινόμενο το λόγο πάρα πολύ σύντομα. Ε, Ένα-δύο λεφτάκια Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συνάντηση. Άρα, έχετε τη σκητάλη για πέντε λεπτά και να προβείτε σε κάποια τελική δήλωση. Merci Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κάποια από τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης είναι τα εξής. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, με βοήθησε να καταλάβω το τι θέλουν από εμένα οι εκπρόσωποι των πολιτών, εάν με ορίσουν ως επίτροπο οι ανησυχίε σας για τον προπολογισμό της πολιτικής συνοχής ε, πράγματι εισακούστηκαν και σας διαβεβαιώ ότι θα τις μεταφέρω στο σώμα των επιτρόπων. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε σημαντικά μηνύματα για το θέμα της ε, συνοχής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και των μεταρρυθμίσεων που είναι θέματα που αγγίζουν το ένα το άλλο, σε βαρές ανησυχίες για την απλοποίηση, ανησυχίες για το γιατί είδους μεταρρυθμίσεις μιλάμε, τι εννοούμε ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, ποιες είναι οι μέθοδοι, για την κλιματική αλλαγή και το σχέδιο δράσης ε, και για την συνεισφορά της πολιτικής συνοχής ε, και την συνεκτικότητά της με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Και αυτό το σημειώνω επίσης για την Ήπεθρο. Οι ανησυχίες ότι υπάρχει μια σύγκληση ε, και βεβαίως οτιδήποτε αναφέρθηκε σε σχέση με τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, ε, η ανησυχία με τον προϋπολογισμό του φύλου σε οτιδήποτε κάνουμε και βεβαίως ε, οι τοπικοί εταίροι και ενδιαφερόμενα μέρη. Όλα αυτά λοιπόν τα σημειώνω, να αναφέρω, ε, ανέφερα τα βασικά σημεία. Ανέφερα επίσης ότι θα είμαστε σε επαφή μαζί σας, ε, αλλά βεβαίως Δεν ανέφερα κάποια άλλα πράγματα. Θα είμαι οπωσδήποτε σε επαφή με την Επιτροπή των Πεφυρίων, την ΕΟΚΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Θα είμαι λοιπόν σε στενή επαφή μαζί τους και με τους διαχειριστές των διαφόρων ταμείων που έχουμε στην Ευρώπη για να δημιουργήσουμε πακέτα τα οποία ε, πραγματικά θα καταστήσουν το σύνολο κάτι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μέρων του. Θα προσπαθήσω να επισκεφθώ όλες τις περιφέρειες τους πρώτους έξι μήνες και βεβαίως ε, και εντός της ε, Κομισιόν θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους. Είναι δύσκολο να έχουμε καλά αποτελέσματα εάν δεν είμαστε σε στενή επαφή με τις μεταφορές, οικονομία, περιβάλλον, δουλειές. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε ως ομάδα και σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε αυτό. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν να προετοιμάσω αυτήν την ε, παρουσίαση τις απαντήσεις μου, ειδικά όσους δουλεύουν στις διάφορες υπηρεσίες και ήταν ε, πολύ υπομονετικοί, πολύ επαγγελματίες και πάντα έτοιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου για να μπορέσω και εγώ να ενημερωθώ, να έρθω μπροστά σας και να προσπαθήσω να απαντήσω επαρκώς στις ερωτήσεις σας. Να ευχαριστήσω και τους Ερμηνείς. Γιατί Βεβαίω, ε, χάρη σε αυτούς ε, συνεννοούμαστε και σας ευχαριστώ όλους. Ε, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και την απόλαυσα. Σας ευχαριστώ. Madame la Κύριε Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, Αυτά τα χειροκροτήματα διερμηνεύσατε τα ως ευχαριστίες εκ μέρους Επιτροπής μας για τις απαντήσεις που δώσατε, στις ερωτήσεις που σας ετέθησαν. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ποιότητα των ερωτήσεων που έθεσαν. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις διαστάσεις και όλες τις πτυχές ώστε τώρα πλέον να μπορέσουμε να προβούμε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητα μαζί με τους συντονιστές για να δούμε κατά πόσον θα σας συγκρίνουμε ως επίτροπο. Έπρεπε να έχουμε αυτή την ακρόαση που ήταν ε, μεγάλης διάρκειας, ποιοτική ιδιαίτερα εξαντλητική, διεξοδική. Οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα στην Επιτροπή μας ε, ήταν πραγματικά πολύ ποιοτικέ, αλλά να μην φλιαρίσω άλλο, παρότι το συνηθίζω, διότι πρέπει να σεβαστούμε τον τύπο που επιβάλλει αυτή τη στιγμή να συνεδριάσουμε μαζί με τους συντονιστές για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση, διεξοδικότατη, ενδελεχέστατη αξιολόγηση των απαντήσεων που μας δώσετε κύριε Φερέρα σε όλες τις ερωτήσεις και όλες τις διαστάσεις και πτυχές της περιφερικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για τους συντονιστές και τους βουλευτές λέω ότι και κλεισμένο των θυρών αύριο το πρωί από τις 10 και τις 12, έως τις 12.30 θα συνεδριάζουμε στο 5ε2 και μετά θα συντάξουμε την γνωμοδότησή μας, την οποία θα απευθύνουμε στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διερμηνείς για την καταπληκτική τους δουλειά. Ευχαριστούμε.